Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε αν θέλετε την απογευματινή μας συνεδρίαση με το σημείο 11 της Μεσσίας Διατάξεως Δημόσια Ακρόαση για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Να καλωσορίσω τους ε, προσκεκλημένους μας ομιλητές Ερικάσορ Μισελ Αλιετά Joshua Ryan Collins να ευχαριστήσω όλους για την παρουσία τους στην ακρόαση αυτή η οποία λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της ε, έκθεσης ε, πρωτοβουλίας για την ίδια χρηματοδότηση της Επιτροπής μας περιμένουμε και το έγγραφο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο. Έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα αυτό, όπως γνωρίζετε. Έχουμε λοιπόν σήμερα την ευκαιρία και τη χαρά να μπορούμε να το συζητήσουμε με διάφορους διακεκριμένους ομιλητές, ιδιαίτερα τον κύριο Αλγίτα, που όχι μόνο στα πλαίσια του κανονισμού αλλά ευρύτερα έχει ασχοληθεί και έχει μελετήσει το θέμα αυτό και μας ενδιαφέρει πολύ να καταλάβουμε πώς εφαρμόζει αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες στο συγκεκριμένο θέμα. Οι ομιλητές έχουν λοιπόν 10 λεπτά για να απευθυνθούν στην Επιτροπή μας και μετά ο εισηγητής και άλλα μέλη βεβαίως θα παρέμβουν. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον κύριο Άσα, τον επικεφαλής του προγράμματος ε, του περιβαλλοντικού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών. Ε, παρακαλώ κύριε Άσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ συνεισηγητά με μεγάλη ικανοποίηση είμαι εδώ σήμερα μαζί σας. Πριν από αρκετά χρόνια στην ε, Σύνοδο του Ρίο το 1992 κάποιοι βασικοί χρηματοπιστωτικοί φορείς είχαν ασχοληθεί με το πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Όλα αυτά κατέληξαν στην πρωτοβουλία UNAP την οποία σας παρουσιάζω σήμερα, UNEP μάλλον. προκειμένου να ενσωματώσουμε θέματα διακυβέρνησης και περιβαλλοντικά από το 2006 με τον κύριο Ανάν στο Παγκόσμιο Σύμφωνο έχουμε σήμερα το 70% των συνυπογραφών των διεθνών θεσμικών επενδυτών κατόπιν με τον πρόεδρο Κιμούν έχουμε το 25% των παγκοσμίων εισφορών στα ασφαλιστικά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Επίσης ε, συνομαδοποιήσαμε τους εκπροσώπους των πιο σημαντικών κεφαλαιογορών του κόσμου μαζί με τις αξιολογήσεις ε, πιστοτικών αποθεματικών. Παρότι έχει σημειωθεί λοιπόν σημαντική πρόοδος εθελοντική περισσότερη από το 1992, η κοινωνία μας είδε αλλαγές που δεν μπορούσαν να την έχουν φανταστεί οι συνειδητέ αυτή τη πρωτοβουλία. Το 2017 ήταν η δεύτερη πιο θερμή χρονιά που, ξε... που έπεται μόνο του 16 με τυφώνες, ε, διάφορες φυσικές καταστροφές, πλημμύρες με εκατοντάδες δισεκατομμυρίων δολαρίων ζημιές και αστικές ευθύνες όχι μόνο συνδεδεμένες με το περιβάλλον και ζημιές και δυσκολία διαχείρισης των φυσικών πόρων. Τον τελευταίο αιώνα ο πλανήτης έχει χάσει 50% των υδάτινων πόρων του και σημαντικό ποσοστό των δασών όπως και των ε, ε, Τέλος πάντων. Χρειαζόμαστε λοιπόν να αλλάξουμε ταχύτητες προς μια... ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνου που θα κοιτάει προς το μέλλον για μια βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία χαμηλή στον άνθρακα και θα πρέπει να διαβρύνουμε το αποθεματικό των επενδύσεων που θα είναι διαθέσιμες για να αντισταθμίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Επομένως η συζήτηση αυτή είναι πολύ επίκαιρη. Το έγγραφο συνοδεύει και το, την αντίστοιχη προσπάθεια της Κίνας ε, για να αν, το χρηματοπιστωτικό αρχιεκτονικό πλαίσιο, ώστε να έχουμε ένα βιώσιμο και υπεύθυνο σύστημα, το οποίο είναι υψή της προτεραιότητας αν είναι να έχουμε μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία. Με αυτήν την εισαγωγή θα ήθελα να σχολιάσω κάποιες από τις συστάσεις για το σχέδιο δράσης ε, της ε, βιώσιμης χρηματοδότησης. Συνολικά θεωρούμε ότι η έκθεση ε, ομαδοποιεί μια σειρά από πολύ σημαντικά πρότυπα που αν υλοποιούντο θα ήταν πραγματικά μια όθηση. Το ακόλουθος σχολιασμός επικεντρώνεται σε κάποια επιμέρους ε, σημεία και δεν συνιστά μια ριζικά διαφορετική τοποθέτηση ή κατεύθυνση. Καταρχάς για το πεδίο εφαρμογή και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Το αρχικό πεδίο συμπεριλαμβάνει παραπομπές ε, σε διάφορους παράγοντες ε, διακυβέρνησης, αλλά όπως ομολογούν και οι συνυπογράφοντες του, η πιο σημαντική συνιστόσα είναι η πράσινη και εντός αυτής το περιβάλλον. Και στην ουσία η, ο μετριασμός των εκπομπών ε, αερίων θερμοκηπίου. η βιώσιμη χρηματοδότηση δεν είναι μόνο εσωτερικό μέσο στα ευρωπαϊκά σύνορα, θα πρέπει να το βλέπει κανεί ως ένα μέσο αντιστάθμισης πιέσεων από το εξωτερικό, μεταναστευτικών, ε, ασφάλειας ε, της ε, προμήθειας των τροφίμων κτλ. Στην χρηματοπιστωτική δομή ε, σημαντικό ρόλο ε, διαδραματίζουν και οι τράπεζες όπως και η κεντρική τράπεζα. Εμείς λοιπόν συνιστούμε ότι είναι σημαντικό για την Ένωση να δει το επίπεδο της φιλοδοξίας που επιθυμεί να ακολουθήσει και οι τράπεζες να, είναι, να συνεργάζονται πιο στενά με την κατεύθυνση αυτή. Τώρα, η ταξονομία προτείνεται είναι αυτό που πιο πολύ πλησιάζει σε μια συνολική αρχή μια δηλαδή αρχή κατάταξης, ξεκινώντας από, το, ε, από την περιβαλλοντική αλλαγή. Δηλαδή να ταυτοποιηθεί ως βιώσιμη συγκεκριμένες δραστηριότητες ή συνδιαλλαγές εντός κάθε οικονομικού πεδίου δραστηριότητας και με τις προσπάθειες της διεύνησης αυτής της κατάταξης θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε ροές εντός των υφισταμένων ή τροποποιημένων ορίων χρηματοδότησης. Αλλά μια τέτοια προσέγγιση θα δυσκολευτεί να παρακολουθήσει τις αλλαγές. Και θα δυσκολευτεί επίσης να εξασφαλίσει ότι θα είναι ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγέτης και θα παρακολουθεί τις εξελίξεις. Στο μέλλον θα εστιαζόμαστε πιο πολύ στον αντίκτυπο, πιο πολύ στην κινητικότητα, στην ενεργειακή απόδοση και όχι στην κατασκευή μονάδων ενέργειας. Ε, το επόμενο βήμα λοιπόν στην ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια πιο ολιστική προσέγγιση ώστε να συμπεριλαμβάνουμε και τον θετικό και τον αρνητικό αντίκτυπο και στους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης. Έτσι θα έχουμε έναν αντίκτυπο πιο κεντρικό με κοινή ορολογία για όλους τους συμμετέχοντες ώστε να εξυπηρετούμε και τον επιχειρηματικό κόσμο και τον χρηματοπιστωτικό κόσμο. Αυτή λοιπόν η χρηματοδότηση του θετικού αντικτύπου είναι μια πολύ θετική έννοια που αναπτύσσει η Κομισιόν και με ικανοποιεί ότι η προσέγγιση αυτή συμπεριλαμβάνεται στο δικό σας σχέδιο για μια συμπερίληψη αυτής της ε, κατάταξης, της μεθοδολογίας. Τότε, από το 2005 όταν είχαμε για πρώτη φορά ασχοληθεί με το θέμα των της ευθύνη των, επενδυτών και των επενδύσεων με υπευθύνους ρυθμιστικών αρχών από διάφορες ε, αρμοδιότητες επί τη βάση του ότι η νομοθεσία σε διάφορες χώρες δεν είναι επαρκώς αφής και ότι χρειάζονται περισσότερες εξηγήσει όταν ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα θέματα τα περιβαλλοντικά. Επομένως τα καθήκοντα των επενδυτών και των καταπιστευματοδόχων είναι απαιτεί αν θέλετε ότι οποιοδήποτε στοιχείο υλικό ή όχι που θα μπορούσε να επηρεάζει την πορεία της επένδυσης θα πρέπει να αναλυθεί από την αρχή και αυτό συμπεριλαμβάνει και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Και παρότι αυτά κωδικοποιούνται όπως το MIFET 2 η έκθεση υπογραμμίζει ότι πρέπει να προσέξουμε κατά πόσον έχουμε αποτυπώσει τα απαραίτητα επίπεδα. Εμείς ενθαρρύνουμε ξεκάθαρα ότι αυτή η ευθύνη θα πρέπει να ενισχυθεί. Υποστηρίζουμε λοιπόν την κατεύθυνση της έκθεσης αυτής και μας ικανοποιεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς τα εμπρός. Η ασφάλιση. Το πυρηνικό τμήμα είναι η διαχείριση του κινδύνου. Ο τριπλός ρόλος της, ε, του κλάδου των ασφαλίσεων είναι η διαχείριση του φυσικού κινδύνου, η χρηματοπιστωτική διαχείριση του κινδύνου και η θεσμική επένδυση. Και εμείς θα θέλαμε να, εμπιστευτούμε, να εστιαστούμε περισσότερο στον θεσμικό επενδυτικό ρόλο τους. Μέσω της ανάλυσης ε, μπορούμε να, μπορεί κανείς να εξασφαλίσει την μείωση ή τον περιορισμό των ζημιών μια οικοσυστημική προσέγγιση και μια προετοιμασία έναντι φυσικών κρίσεων μέσω της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να ενισχύσει το σύστημά της ε, για τις αναλύσεις σεναρίου και την διαχείριση δυνητικών φυσικών καταστροφών. Επίσης, απορροφώντας ε, τα χρηματοπιστωτικά ε, κρούσματα που προέρχονται από φυσικές καταστροφές, κρίσεις και άλλες κινήσεις της οικονομίας μπορούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις επίσης να συνεισφέρουν όπως και στην ενεργειακή απόδοση, την ανάχρηση των κτηρίων και την μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία. Πρέπει πάντως να, αναπτύξουμε παγκόσμιες κατευθύνσεις που είναι η διαδικασία της αξιολόγησης ε, του ασφαλιστικού κινδύνου για όλους τους κλάδους ε, της ε, δραστηριότητας ασφαλιστικής. Θα πρέπει να δούμε τους ρόλους των ασφαλιστικών φορέων που, που μπορούν να συνεισφέρουν δηλαδή προς τη μετάβηση σε μια πρώτη βιώσιμη και πιο πράσινη οικονομία. Σχεδόν έχω τελειώσει λέει ο μιλητής ο οποίος ομιλεί με την ταχύτητα του φωτός. Τώρα, αυτά που συνιστούν την προσδοκία και των επιχειρήσεων και των θεσμικών φορέων για την σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η προσαρμογή στα UNGP, δηλαδή κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και οι επενδυτές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να δουν τι σημαίνουν για αυτούς οι UNGP αυτές κατευθυντήριες γραμμές στην πράξη ώστε να αναπτυχθούν ε, πλαίσια πολιτικής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, αποφεύγοντας ε, τον κατακαιρματισμό και τα αναμειγμένα μηνύματα προς τον κλάδο. Για την βιώσιμη υποδομή πρέπει να μειωθούν κατά τρία τέταρτα οι εκπομπές ε, αερίων θερμοκηπίου με το 2050, με συγχωρείτε, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το έργο και του ΙΦΙΚ και με πολύ μεγάλη χαρά βλέπω σήμερα τους εκπροσώπους του ΙΦΙΚ εδώ σήμερα κυρίως λόγω του μικρού μεγέθους συγκεκριμένων επενδυτικών έργων υπάρχουν ομοιότητες ε, με, τις, ε, με τα έργα μεγαλύτερης υποδομής ως προς την δηλαδή πτυχή την λογοδοσία που αναλαμβάνεται ή το ρίσκο που αναλαμβάνεται από τα έργα αυτά σχετικά με, τις, ε, με την προετοιμασία κλιματικών φαινομένων. Η ενεργειακή απόδοση και η βιώσιμη υποδομή και εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πιο ρητή ώστε να μην είναι ε, απλώς μια αναφορά στιγμιαία, αλλά είναι μια συνεχής διαδικασία που να επιτρέπει την κατάλληλη χρηματοδότηση των ροών αυτών. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν ε, στοιχεία που είναι συγκεκριμένα για τα κτίρια ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο το δυναμικό των έργων αυτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα περνάμε στον Επιστημονικό Σύμβουλο του Κέντρου Διεθνών Μελετών και Προβλέψεων, τον κύριο Αλιέτα. Με ένα αρκετά μακροσκελές και σχετικό βιογραφικό. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που με καλέσατε στην ακρόαση. Ε, επειδή υπάρχει τερμηνία θα μιλήσω γαλλικά για να εκφραστώ καλύτερα για ένα δύσκολο θέμα. Ε, Στα γαλλικά θα σταθώ σε δύο σημεία όσον αφορά την πολιτική οικονομία. Πρώτα πρώτα η πολιτική ευθύνη, τα χρηματοοικονομικά να μπορέσουν να υπερβούν την τραγωδία. Και από την μεριά είναι τα μακροοικονομικά όσον αφορά το μετασχηματισμό των δομών παραγωγής και κατανάλωσης για βιώσιμη ανάπτυξη. Τραγωδία είναι το συλλογικό ρίσκο πέραν αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις του ορίζοντος ας πούμε. Το ρίσκο προέρχεται από κάποιο είδου ε, εγγενή ανασφάλεια όσον αφορά την αξιολόγηση του ρίσκου και όσον αφορά τις επενδύσεις. Αυτή η βεβαιότητα αλλάζει κατά τρεις τρόπους στην πολιτική. Πρώτα-πρώτα η ζημιά από το κλίμα, και η προβλή του κέρδους είναι αλληλένδετα και έτσι έχουμε μεθόδους ασφάλειας διαφορετικές σε σχέση με την σημερινή παγκοσμιοποίηση. Οι τρόποι αξιολόγηση του κινδύνου δεν είναι επομένω οι ίδιοι. Άρα αυτή η τραγωδία σημαίνει συνέχεια των προτεραιοτήτων της πολιτικής πέραν της προεκλογικής περίοδου. Επίσης, η διασυνοριακή υπερεθνική συνεργασία είναι απαραίτητη, ούτω ώστε να είναι βάση οι νέες τεχνολογίες προς του περιβάλλοντος. Επομένως, μια πολιτική συμφωνία είναι αν απαραίτητη στην Ένωση πέραν των μικροκομματικών συμφερόντων πέρασε μια τριακονταετία ούτως ώστε να υπάρχουν εγγύησει για να υπάρξουν οι, το, το κατάλληλοι λοιπόν πόροι. Και τι χρειάζεται. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες για τις επενδύσεις. Και αυτό είναι η έννοια της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Αυτά με τη στήριξη του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού με επιπλέον ιδίους πόρους και ίσως αυτή που στεμένει αξία μπορεί να παραγάγει κάτι σε επίπεδο ένωσης με την επικουρικότητα. Αυτό που δεν μπορεί να καταφέρει μόνο της κάθε χώρα. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από το win-win. Να πως πρέπει να αντιληφθούμε τις επενδύσεις. Γι' αυτό μιλάω για θωράκιση του προϋπολογισμού με νέου είδους ιδίους πόρους σε σχέση με τις προτεραιότητες που θα τάξουμε. Δούμε τώρα ποια είναι τα σχετικά εργαλεία, τα μέσα και ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές, οι βασικοί. Είναι θέμα φορολόγησης του άνθρακα. Δεν είναι τόσο απλό όμως αυτό. Ιδίως αν κοιτάξει κανείς τις παραδοσιακές οικονομίες. Έτσι θα έχουμε λιγότερη ένταση στη χρήση του άνθρακα και επίσης θα βοηθήσουμε την καινοτομία. Όμως υπάρχουν διάφορες επιλογές. Πρώτα-πρώτα ο φως για τον άνθρακα, γνωστός, δίνει πόλου στην κυβέρνηση, καλό αυτό. Αλλά δεν παρέχει εγγυήσει όσον αφορά την μείωση των εκπομπών σε συγκεκριμένη βάση. Cap and trade. Το μειονέκτημα είναι η τιμή όπως έχει διαπιστωθεί εδώ και κάποια χρόνια. Επομένως, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον υπάρχει κάποιο είδους ε, όριο στην ε, τιμή. Άρα έτσι να φύγεται ο Ριπένων και όλα αυτά ανάλογα με το τι γίνεται. Ούτω ώστε να μπορεί να συνεχιστεί η εξέλιξη της οικονομίας. Και έτσι να κάνουμε τη σχετική προσαρμογή των ορίων της μόλυνσης. Τώρα η θεωρητική τιμή όσον αφορά τις δραστηριότητες. Shadow price. Αυτό ενσωματώνεται στις επενδύσεις έτσι έχουμε πράσινες επενδύσεις. Και ο φόρος για τον άνθρακα, η τιμή για τον άνθρακα και το κόστος της κατεδάφισης θα πρέπει να καλυφθεί και έτσι καταλήγουμε στη θεωρητική τιμή και αυτά, αυτά τα μεγέθη θα πρέπει να συγκλίνουν. Και αυτό μας δείχνει ότι θα πρέπει αυτοί οι παράγοντες να συνδυαστούν. Επίσης, η αλλαγή στα χρηματοοικονομικά, ούτω ώστε να υπάρχει καινοτομία για τα μεγάλα έργα υποδομής. Οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί έχουν το εξή πρόβλημα. Θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ε, στρεβλώσεις. Άρα θα πρέπει να καλυφθεί και αυτή η έκπτωση όσον αφορά τον άνθρακα και να υπάρξουν αντίστοιχες επενδύσεις. Να υπάρχει συντονισμός για τους εξωτερικούς παράγοντες και επίσης αξιοποίηση από τις αγορές. Άρα καλύτερη υγεία, λιγότερη μόλυνση και επιτυχίες και στο μέτωπο της ενέργειας. Όλα αυτά να μπορεί να τα αξιοποιήσει η αγορά. Και όλοι αυτοί οι παράγοντες, οι εμπλεκόμενοι, παίζουν σημαντικό ρόλο. Οι κρατικές τράπεζες, οι κρατικοί επενδυτές μπορούν να χρηματοδοτήσουν μακρόπνο έργα. Είναι επομένω οι επενδυτές οι οποίοι θεσμικά είναι οι υπεύθυνοι για την διακυβέρνηση των επιχειρήσεων λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του στρατηγικούς βιώσιμης ανάπτυξης και οι κεντρικές τράπεζες πρέπει τις υποχρεώσεις για το περιβάλλον τους λάβουν υπόψη στην πολιτική τους. Χωρίς κεντρικές τράπεζες δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες δραστηριότητες. Δύο λόγια τώρα, μια που έχω το χρόνο, όσον αφορά τις μακροοικονομικές πολιτικές. Προσωμιώσεις με κάποια μοντέλα πέρα από το Nordhaus. Και έτσι εδώ ενσωματώνουμε και τον ρόλο αυτών των οικονομικών παραγόντων. Και έτσι να είναι ομαλή η ενεργειακή μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία παρά το ότι είναι σίγουρο θα υπάρξουν ζημίες και τεχνολογική διαφορά σε σχέση με τις εκπομπές του άνθρακα. Τρία πράγματα πρέπει εδώ να συνδυαστούν τουλάχιστον όσον αφορά αυτές τις προσημειώσεις η φορολόγηση του άνθρακα, οι επιδοτήσεις όσον αφορά τις πράσινες ε, και το πράσινο επιτόκιο, ούτως ώστε να δοθούν κίνητρα σε αυτές τις επενδύσεις που θέλουμε να υπάρξουν. Και γίνεται αυτή η προσωμείωση λαμβάνοντας υπόψη όχι τις απλές ζημίες όπως το North αλλά πολύ πιο μεγάλη ποικιλία ζημιών. Επομένως θα πρέπει να είναι υψηλός ο φόρος για να αποθαρρύνει τις μολύνουσες τεχνολογίες μειονέκτημα είναι το ότι οι επενδυτές που επενδύουν σε τέτοιες πράσινες επιχείρησεις έχουν ζημίες και αυτές μπορεί να είναι πολύ σημαντικές οι ζημίες γιατί πια τα στοιχεία ενεργειακού ενεργητικού δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Επομένως έχουμε δυνάμεις σε πολιτικό επίπεδο που αντιδρούν. Άρα προσκρούει εκεί πέρα ο φόρος του άνθρακα, συν οι επιδοτήσεις. Οπότε μπορεί να μειωθεί αυτός, να είναι πιο ομαλή, πιο ήπια η εφαρμογή του. Και ε, προστίθεται ένα δεύτερο εργαλείο για τις επενδύσεις που δεν ε, έχουν άνθρακα. Σύμφωνα με την κοινωνική αξία των εκπτώσεων. Οπότε έτσι μπορούμε να υποστήξουμε τις επενδύσεις και έτσι δεν προβαίνουμε στην αξιολόγηση των εταιριών, των... αυτό που μπορεί παίρνει τέλο πάντων. Εάν επομένω επιβραδύνουμε την μετάβαση, μπορεί να προκύψει κάποιο είδου παρέκκληση από αυτή τη διαδρομή των δύο βαθμών. Επομένως, φόρος συν πράσινο επιτόκιο, συν επενδύσεις, τότε βελτιώνουμε με περισσότερα κέρδη την υπόθεση αυτή και ως αποτέλεσμα έχουμε κάτι ενδιαφέρον γιατί τότε είναι δυνατόν να έχουμε μια μετάβαση με περισσότερα κέρδη και το χρηματοοικονομικό σύστημα παραμένει σταθερό φροντίζει το επιτόκιο κεντρική τράπεζα δίνοντας μία εγγύηση σε αυτά τα πράσινα ομόλογα. Δεν μπορούμε να έχουμε ενεργητικό χωρίς τέτοιου είδους φροντίδα. Και μόνο στη μακροοικονομική της πολιτική θα το κάνει αυτό η κεντρική τράπεζα για τον πράσινο κλάδο. Οπότε έτσι παρέχει εγγύσεις, πιο ποιοτικέ. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ράιον Κόλλιν. Ε, ερευνητής στο Ινστιτούτο Καινοδομίας ε, και Κοινοφιλών Σκοπών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την μόλι Σκοτ Κέιτο που με κάλεσε σήμερα εδώ. Εγώ θα εστιάσω στον τραπεζικό τομέα και τον ρόλο της νομισματικής πολιτικής ε, και της ε, ρύθμισης ε, που είναι ο τομέας επί το οποίο εργάζομαι τα τελευταία δέκα χρόνια στο νέο Ίδρυμα περί οικονομικών στο Λονδίνο. Πρώτα απ' όλα Έχουμε το μέγεθος της πρόκλησης ε, που αντιμετωπίζουμε. Η έκθεση Άσλογκου μιλάει για 170 δισεκατομμύρια το χρόνο, ένα κενό χρηματοδοτικό για το κλίμα. Μιλάμε για κάτι το τεράστιο. Και η έκθεση σωστά επισημαίνει ότι δεν αρκεί να βασιζόμαστε στον δημόσιο τομέα. Πρέπει να κινητοποιήσουμε τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Εντός αυτού του τομέα ε, υπάρχουν ε, πάνω από ε, έναν δύο παίκτες και χρηματαγορές και ο Έρικ νομίζω το υπογράμμισε. Το πρώτο το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι οι κεφαλαιαγορές και τα κράτη όταν δαπανούν ή επενδύουν, επενδύουν υφιστάμενα χρήματα. Δηλαδή από κάπου αλλού τα παίρνουν πριν τα ξοδεύσουν. Αντιθέτως, οι εμπορικές τράπεζες και οι κεντρικές τράπεζες όταν δαπανούν μπορούν να δημιουργήσουν ε, νέο χρήμα, νέα αγοραστική δύναμη μέσω του δανεισμού, της πίστης και της δημιουργίας πίστης, γιατί όταν δανείζουμε δίνουμε κάτι. Οπότε οι τράπεζες δημιουργούν ε, πίστοση γύρω στο 97% όλων των νέων χρημάτων στην οικονομία και για να αντιμετωπίσουμε το μέγεθος αυτής της μετάβασης αυτό νομίζω είναι το βασικό γεγονό που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Δυστυχώς ε, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι το τραπεζικό σύστημα ως έχει αυτή τη στιγμή μπορεί να ανταποκριθεί. Αυτό εν μέρη γιατί η κλιματική αλλαγή είναι μια περίπλοκη διαδικασία και ο αντίκτυπος της είναι απρόβλεπτος Υπάρχουν πολλά μη γραμμικά στοιχεία. Υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει κάποιο στοιχείο καμπής ε, πέρα από το οποίο οι μόνοι υπάγοι θα λιώσουν και θα απελευθερώσουν μεθάνιο αλλά είναι δύσκολο να προβλεφθεί κάτι τέτοιο οπότε δεν μπορεί να ενταχθεί σε παραδοσιακές αγορές οι οποίες λειτουργούν σε ένα χρονικό πλαίσιο ενός έως πέντε ετών και Ήδη αυτό το έφερε και ο Μισελ. Υπάρχει λοιπόν ε, μια συστημική λάθος τιμολόγηση αυτών των ζητημάτων. Όπως είπε ο Νίκολας Στέν για τη μεγαλύτερη αποτυχία της αγοράς ε, στον κόσμο. Το θέμα είναι το τι κάνουμε λοιπόν. Πολλές από τις ε, συνεισφορές λοιπόν στην έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικές, οπωσδήποτε η κατηγοριοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική και οι δράσεις οι οποίες προτείνονται επίσης στο σχετικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ θετικέ. Αλλά αυτό το οποίο δεν βλέπω εγώ στην έκθεση είναι τα διαρθρωτικά ζητήματα. Το πώς δηλαδή θα καταφέρουμε το τραπεζικό σύστημα να στηρίξει την μετάβαση. Νομίζω ότι ο χρόνος της εθελοντικής αποκαλύψεως ε, σιγά σιγά θα πρέπει να τελειώσει, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε πια σε θελοντική αποκάλυψη για τα στοιχεία ενεργητικού που αφορούν ε, βιομηχανίες ε, του άνθρακα. Έχουμε πάρα πολλά ε, εργαλεία τα οποία αγνοεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας και δεν υπάρχει λόγος να θεωρούμε ότι επειδή οι ρυθμιστικές αρχές ή οι κεντρικές τράπεζες ζητάνε τώρα να υπάρξει εθελοντική αποκάλυψη ότι θα γίνει αυτό. Πρέπει, θεωρώ εγώ λοιπόν ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική αυτή η αποκάλυψη. Πρέπει όμως να πάμε ακόμη παραπέρα. Ένα από τα βασικά διδάγματα της οικονομικής κρίσης ήταν ότι η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών ότι αν τις αφήσουμε δηλαδή να κάνουν τη δουλειά τους θα κάνουν τις βέλτιστες επιλογές δεν είναι πλέον ε, αξιόπιστοι και είναι σαφές ότι αν αφήσουμε τις τράπεζες μόνες τους να αναπτύξουν μόνες τους τα δικά τους κριτήρια κινδύνου έχουν την τάση να οδηγούνται σε κερδοσκοπικές ε, φούσκες έξω και αυτό το οποίο αναπτύχθηκε ως μακροπροληπτική πολιτική κάποιες τράπεζες έχουν μια ξεκάθαρη εντολή όπως η Τράπεζα της Αγγλίας Βεβαίω στην Ευρώπη υπάρχει ένα διαφορετικό φορέας, αλλά ο στόχος της μακροπροληπτική πολιτικής είναι ακριβώς να εξετάζουν τον συστημικό κίνδυνο. Και ένας βασικός τομέας που επισημάνθηκε μετά την κρίση ήταν η αγορά των ακινήτων. Πριν από την κρίση, αν προσπαθούσαμε να πείσουμε τους κεντρικούς τραπεζίτες να έχουν οι τράπεζες περισσότερο κεφάλαιο σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια θα έλεγαν ότι δεν ξέρουμε πόσο είναι ο κίνδυνος, δεν είναι φούσκα, καλύτερο είναι να ξεκαθαρίσουμε μετά τα πράγματα. Βεβαίως τώρα εκ των υστέρων είναι προβληματική αυτή η άποψη. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι ο κίνδυνος της μετάβασης της ε, κλιματικής αλλαγής είναι ένας τέτοιος κίνδυνος και δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε μεμονωμένες τράπεζες ή στη μακροπροληπτική πολιτική των τραπεζών για ε, τέτοιους μακροοικονομικούς κινδύνους που αφορούν ολόκληρο το σύστημα. Χρειάζεται λοιπόν μια προληπτική παρέμβαση, κάτι το οποίο κάνει η μακροπροληπτική πολιτική. Βλέπουμε τώρα ότι η κεντρικές τράπεζες αναγκάζουν τις ε, εμπορικές τράπεζες να διακρατήσουν μεγαλύτερο ποσοστό κεφαλαίου σε σχέση με ορισμένους κλάδους, ε, χαρακτηριστικά είναι τα στεγαστικά δάνεια και σε άλλους κλάδους και από ό,τι φαίνεται αυτό λειτουργεί. Στην Ελβετία φαίνεται ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της εφαρμογής αυξημένης πίστης και μείωσης στον ε, δανεισμό για στεγαστικά δάνεια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν πρέπει να το πάρει σοβαρά αυτό και να σκεφτεί να ανεβάσει το στο κεφαλαίου ή άλλες μορφές ε, κατεύθυνσης της ε, πίστης για να στηρίξει τις πράσινες επενδύσεις και να μειώσει τις επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα. Γιατί έτσι μετά υπάρχει ακριβώς ένας εγκλωβισμός σε αυτές τις ε, τεχνολογίες. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι βεβαίως, ε, πέρα από το να αναγκάσουμε τις τράπεζες. Μπορούμε να έχουμε αντικυκλικά αποθέματα, Και βεβαίως υπάρχουν, υπάρχει και η πράσινη πίστη Είχαμε κάτι ανάλογο στη μεταβολημική περίοδο για την κατεύθυνση της πίστης στην Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο για να στηριχθούν στρατηγικοί τομείς της οικονομίας οπότε ουσιαστικά απαιτούμε από τις τράπεζες να έχουν ένα 30% του ισολογισμού σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Η Ινδία το κάνει αυτό αυτή τη στιγμή για τον δανεισμό για τις ΑΠΕ κατά προτεραιότητα το οποίο εφαρμόζει η Κεντρική Τράπεζα. Νομίζω καλό θα ήταν ε, το σχέδιο δράσης να εξετάσει ακριβώς ε, την κατεύθυνση της ε, πίστης. Βεβαίως εναλλακτική θα ήταν να έχουν οι τράπεζες λιγότερο κεφάλαιο αρκεί να δίνουν περισσότερα πράσινα δανεία. Είναι καλή ιδέα αλλά λάθος μέσο γιατί έτσι υπονομεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα για να υπάρχει περισσότερη πίστη στα κατάλληλα τμήματα της οικονομίας. Οπότε εγώ θα ήμουν υπέρ ενός παράγοντα ο θα τιμωρούσε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Να μιλήσω τώρα γενικότερα για την νομισματική πολιτική και εδώ πέρα ήταν απογοητευτική η έκθεση καθώς δεν αναφέρθηκε ο ρόλος της νομισματικής πολιτικής αυτό είναι προβληματικό. Ε, το πιο προφανές εδώ είναι ότι η ΕΚΤ δημιουργεί 60 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε μήνα αυτή τη στιγμή, κατά το οποίο επηρεάζει πολύ την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά δυστυχώς τα κριτήρια εφορίας δεν περιλαμβάνονται στα κριτήρια της ε, τράπεζας. Αυτό το οποίο θα έλεγα εγώ λοιπόν, ότι η ουδετερότητα της αγοράς δεν είναι το ίδιο με την αηφορία ή η ουδετερότητα για την κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν, υπάρχει έρευνα το London School of Economics που λέει ότι οι αγορές ε, της ΕΚΤ ε, ουσιαστικά στηρίζουν ε, κλάδους με υψηλό, υψηλές εκπομπές γιατί ουσιαστικά αγοράζουν εταιρικά ομόλογα το πρόγραμμα αυτό το ESPP Κάτι το οποίο βεβαίως ε, είναι διακριτική μεταχείριση ει βάρο των μικρότερων εταιριών ε, που κατά πάσα πιθανότητα θα καινοτομήσουν στον πράσινο τομέα. Πρέπει λοιπόν να το δούμε αυτό. Και η έκκλησή μου προ την ΕΚΤ είναι να αναλάβει ηγετικό ρόλο εδώ πέρα ενθαρρύνοντας τις ε, τράπεζες να αποκαλύψουν τον κλιματικό κίνδυνο. Αλλά πρέπει και η ΕΚΤ να κάνει το ίδιο στον ισολογισμό της και σε σχέση και με τις εγγυήσει ε, που απαιτεί όταν δίνει δάνεια σε τράπεζες. Και έτσι θα δώσει το παράδειγμα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για τις τοποθετήσεις σας. θα διαφωνούσα με αυτόν τον υποστηρικτικό παράσινο παράγοντα γιατί οι εναλλακτικέ προς την ποσοτική χαλάρωση θα άφηναν τα πράγματα όπως έχουν. Τα οποία και πάλι θα οδηγούσαν σε χρηματοπιστωτική αστάθεια. Μια μετριασμένη λοιπόν υποστήριξη δεν θα έπρεπε να αποκλείεται τόσο εύκολα, λέει ο πρόεδρος. και με ικανοποίησε πολύ και το οργανικό μείγμα μέτρων που πρότεινε ο καθηγητής Αλιετά. Εν αυτό ήταν εν είδη σύντομου σχολείου από πλευρά. μου. Θα ακούσουμε βεβαίως ε, τον συγκητή και στους σκιώδη. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Φέρμπερ. Η Μόλι πρώτα έχει το λόγο και μετά ο κύριος Φέρμπερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους τρεις ομιλητές. Είναι τεράστιο το μέγεθος της εμπειρογνωμοσύνης που είναι παρούσα στην αίθουσα αυτή τη στιγμή. Και εγώ προσπάθησα να καλύψω κάποια από τα πολλά και διάφορα θέματα που κανονικά συμπεριλαμβάνει το πεδίο αυτό της ε, σύντομης δικής μου έκθεσης για τα κλιματικά, για τις επενδύσεις ε, και τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα και λιγότερο για το τραπεζικό. Εγώ νομίζω ότι η, η κατάταξη που προτείνεται στην έκθεση θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι θα μπορούσε κανείς να υιοθετήσει μια ακόμα πιο συγκεκριμένη κατάξη. Βέβαια το πρόβλημα είναι με μια σταθερή ταξονομία να υποστηρίξει κανείς τη μεταβατική περίοδο, να την διαβεί. Αυτές η δυναμική ορολογία θα μπορούσε να δίνει μια διέξοδο. Μεταξύ των υπολείπων και εγώ εξετάζω και θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε στο τελευταίο τμήμα της εντολής μας ε, την ε, ε, φορολόγηση του άνθρακα όπως και τις κατευθυντήριες γραμμές της πίστοσης την οποία παραχωρεί και η Κεντρική Τράπεζα δηλαδή. Αλλά θα εστιαστώ κυρίως σε αυτό την, την διαχείριση του κινδύνου και το σχετισμό με, τις, ε, με τον κλάδο των ασφαλίσεων. Ότι δηλαδή δεν κάνουμε όσα μπορούμε ως διαχειριστές κινδύνου, αλλά βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει κανείς αυτό όταν μιλούμε για έλλειψη προβλεψιμότητας. Στη γεωργία έχουμε εστιαστεί σε έναν τομέα που δεν έχουμε επαρκώς ε, αναλύσει και διαχειριστεί τον κίνδυνο ιδιαίτερα σε σχέση με τις τιμές ε, και του εδάφους και των λιπασμάτων και του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής. Σε περίπτωση που αυξηθούν ακόμα περισσότερο οι περιβαλλοντικές πιέσεις, πώς θα θεωρούσατε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί ή το αποτύπωμα του κινδύνου που αναλύεται. Επίσης, ο κ. Κόλλινς μίλησε για την ΕΚΤ, αλλά κανείς δεν αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία ε, φέτος ε, ήταν αντικείμενο μιας επανεξέτασης ε, πρόσφατα δάνεισαν στην, στον αγωγό της Αδριατικής το οποίο έχει πολλά ερωτηματικά βρίσκω Νομίζω ότι στο μέλλον θα έπρεπε να έχουμε συμφωνίε μόνο επί τη βάση τη συμφωνία του Παρισίου, δηλαδή χωρίς ορυκτά καύσιμα, αλλά θα ήθελα και τη δική σα άποψη από αυτού. Uh, ευχαριστούμε. Ο επόμενος. Κύριε Πιετικάνη, σας ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και εμπλουτίζουν την έκθεσή μας. Για παράδειγμα, βλέπουμε πώς ε, αυτό το ενεργητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις τράπεζες. Εμένα με απασχολεί το εξή όσον αφορά αυτή την πρόταση. Αυτή η κατηγοριοποίηση για τον πράσινο φόρο μπορεί η πράσινη επένδυση να είναι πάρα πολύ πράσινη Επίσης όμως μπορεί οικονομικά να είναι πάρα πολύ υψοκίνδυνη ή μπορεί να καταλήξει σε πάρα πολύ κακή διαχείριση. Άρα δεν μου αρέσει αυτή η τακτική των πρασίνων επενδύσεων γιατί τελικά θα πρέπει να υπάρχει και εδώ βιωσιμότητα. Οπότε θα πρέπει στην κατηγοριοποίηση να δούμε ε, βέβαια ε, την πρόταση αυτή σε αντιπαράθεση με το να μην υπάρχει καθόλου φορολογική. <clears throat> Τώρα για να δούμε τους δείκτες. Έχουμε τις εκπομπές του διοξιδίου, έχουμε την ανάλωση ε, των βιώσιμων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οπότε αυτό είναι κάτι δεδομένο. Και υπάρχει ένας κύκλος διάρκειας για τα οικοσυστήματα. Άρα θα πρέπει αυτοί οι δείκτες πρώτα να αποφασιστούν όπως και στον υπολογισμό, στη λογιστική και να δούμε τελικά το πρασίνισμα και η σχετική ετικέτα πώς θα διαμορφωθεί και τι γίνεται με τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα. Άρα είναι θέμα του πώς θα ορίσουμε το πράσινο και το πρασίνισμα. Άκουσα τι είπατε για τον ε, φόρο του άνθρακα, αλλά για πέστε μου τη γνώμη σας για τους ε, δείκτες. Τι άλλα εργαλεία μπορεί να μετέλθετε για να δείτε πού δεν πάει καλά η αγορά σε σχέση με το ποιο είναι το κόστος του να μην κάνουμε τίποτα νομοθετικά. Πολτάνκα. Ευχαριστούμε τους ομιλητές. Είναι πάρα πολύ θετικά τα όσα συζητούμε. γιατί ήρθε η ώρα και, και αργήσαμε κιόλας να συζητήσουμε τι είναι η βιώσιμη χρηματοδότηση. Καθυστέρησε η νομοθεσία, καθυστέρησαν οι εμπλεκόμενοι στα χρηματοοικονομικά. Άρα, λαμβάνουμε υπόψη το τι είπε η ομάδα υψηλού επίπεδου των ειδικών. Επίσης, είναι δύσκολο το θέμα. Γιατί πρόκειται πρώτη κάτι είναι εξελίξη. Άρα να φτιάξουμε ένα πλαίσιο και να το συμπληρώσουμε. Να το γεμίσουμε το ΣΥΠΗΝ. Συγκεκριμένα και συνεχώς. Και με προβληματίζει το ότι η κατηγοριοποίηση αυτή είναι μια αφετηρία. Καλή. Αλλά θα πρέπει παράλληλα να μιλήσουμε για την αποκάλυψη και για τις επενδύσεις. Να μην κάνουμε αυτή την κατηγοριοποίηση και να κάτσουμε να περιμένουμε τα αποτελέσματα. Τέτοια προσέγγιση λέμε που θα αποβεί πιο αξιόπιστη και πιο αποτελεσματική για το μέλλον. Επίσης, άκουσα από τουλάχιστον δύο από τους ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πώς τα κίνητρα είναι τα πιο δόκιμα. Για πέστε μας, ορθώς εφαρμόζονται αυτά τα κίνητρα για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στην αλλαγή που θέλουμε να επιφέρουμε. Ο φόρος αυτός, ο καφέ, Εντάξει, υπάρχει, αλλά είναι αυτό μια αφετηρία επίση. Όμω είναι δεδομένη η κίνδυνη. Όσον αφορά έναν ισολογισμό χρηματοπιστωτικού ιδρύματος πρέπει να δούμε πώς ε, η κίνδυνη αυτή θα είναι σαφής γνωστή και έτσι να δούμε πώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα μπορέσουν να καταλήξουν σε αποφάσεις για επένδυση. Άρα να δούμε τι άλλες προτάσεις θα υποβληθούν. Ε, ευχαριστώ. Η επόμενη συνάδελφος. σας ευχαριστήσω εξαιρετική αυτή η παρέμβαση. Οι συστάσεις της ομάδας εργασίες υψηλού επίπεδου βασίζονται σε θελοντικά μέτρα για να συλλέξουμε ακριβώς δεδομένα για το πώς θα λειτουργήσουν. Θεωρείται ότι οι συστάσεις αυτές που βασίζονται σε θελοντικά μέτρα επαρκούν για να αλλάξουν τα κίνητρα των χρηματαγορών για να κατευθύνουμε επενδύσεις σε πιο βιώσιμους στόχους. Η δεύτερη μου ερώτηση σχετίζεται με την ομοθεσία περιφερειγκαιότητας. Η ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου προσφέρει εξαιρέσεις για τα πράσινα προϊόντα αλλά αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι το πώς τιμολογούμε τους ε, κινδύνους δεν υπάρχει ο κίνδυνος ε, αν εφαρμόσουμε χαλαρά κριτήρια σε όλους ε, να έχουμε ακόμα σοβαρότερα προβλήματα. Σας ευχαριστώ. Λίευε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι, σας ευχαριστώ. Μια ερώτηση έχω βασικά οι επενδυτές ε, πάντα σχεδόν κοιτάνε την απόδοση. Πώς ε, θα φροντίσουμε η απόδοση αυτή να είναι υψηλότερη στα βιώσιμα προϊόντα. Αυτό μπορεί να γίνει βεβαίως αυξάνοντας την απόδοση. Και πώς θα το κάνουμε αυτό διασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους ενδιαφερόμενους ε, χωρίς να αποσταθεροποιήσουμε τις ε, χρηματοφόρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ο Δημήτρης είναι τελευταίος. Θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσες τις τοποθετήσεις που ακούσαμε ε, γιατί τροφοδοτούν μια συζήτηση που για να είμαστε ειλικρινείς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αργήσει να ανοίξει και πρέπει να την εντείνουμε και να τη βαθύνουμε αυτή τη συζήτηση υπάρχουν χώρες όπως η Ινδία ή η Κίνα που κάνουν προσπάθειες σε αυτό το τομέα με εντυπωσιακού ρυθμούς. Πριν από λίγες εβδομάδες ε, διεπίστωσα ότι η Κίνα έχει ξεπεράσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επενδύσεις που κάνει στην καινοτομία και την έρευνα. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτές οι εισηγήσει που κινούνται πέρα από το business as usual ε, μας βοηθάνε πάρα πολύ και θα ήθελα να εμπλουτίσουμε την έκθεση που ήδη είναι σε πολύ καλή κατεύθυνση που έχει ετοιμάσει η συνάδελφος μόλις κότς κάτω, ε, αξιοποιώντας και αυτό το υλικό. Ε, προσωπικά δίνω ιδιαίτερη σημασία στο ταξόνομι, όπως επίσης και στην ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας και της διάχυσης πληροφοριών. Συμφωνώ με την πρόταση για υποχρεωτική διάχυση πληροφοριών γιατί η παραμονή στη ρήτρα της εθελοντικότητας δεν έχει δώσει μέχρι τώρα ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η ερώτησή μου είναι μία. Αν μπορείτε να μας δώσετε ε, περισσότερα στοιχεία, τι να περιμένουμε από το Action Plan ε, το Μάρτιο. Θα έχετε δηλαδή έτσι μια πιο καθαρή δομημένη πορεία να περιγράφεται στο τι και πώς πρέπει να γίνει, βήματα, milestone, στόχους μέσα ή θα μείνουμε σε, πολύ γενικότητες στην περιγραφή. Γιατί το action plan σαν όρος είναι φιλόδοξος και σημαίνει σχέδιο για δράση. Θα έχουμε ένα σχέδιο για δράση το Μάρτιο. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βλέπω κάποιον άλλον να ζητάει το κετσιά εκτός από μένα. Μόλι αν συμφωνείς καθώς το επόμενο θέμα είναι δική σου έκθεση να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο. Λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν, στους ε, προσκεκλημένους μας. Τρία-τέσσερα λεπτά το πολύ, αν συμφωνείτε, για να μην χάσουμε πολύ χρόνο. Ποιος θα ξεκινήσει. Ναι. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος να απαντήσω σε ερωτήσεις που μπορώ να απαντήσω. Άκουσα τις ε, απόψεις ε, για το θέμα αυτό της ε, κατηγοριοποίησης. Πρέπει να υπάρξει ακριβώς ένας έξυπνος τρόπος να γίνει αυτό, να έχουμε την δυνατότητα να ταυτοποιήσουμε ποιο είναι το σωστό είδος εταιρεία αντί να τα περιμένουμε όλα από τον κατάλογο. Για την εισηγήτρια για τους διαχειριστές κινδύνου και τις ασφαλιστικές εταιρείε. μία από τις προκλήσεις είναι ότι οι διαχειριστές κινδύνου κατά κανόνα ανατιμούν τον κίνδυνο ετησίως και δεν κοιτάνε μακροπρόθεσμα γιατί αν αποδειχθεί μεγαλύτερος ο κίνδυνος μπορούν να αναπροσαρμόσουν τις ε, τιμές. Οπότε θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε και στην ασφάλεια αυτό το οποίο υπάρχει στις ε, επενδύσεις, την ευθύνη δηλαδή των ασφαλιστών να δρουν προς το συμφέρον των πελατών τους και να αντιλαμβάνονται τις μακροπρόθεσμες ε, προοπτικές, παραδείγματος χάρη της γεωργίας δηλαδή όπως υπάρχει ένα σχετικό καθήκον στις επιχειρήσεις. Λοιπόν, για τα κράτη, τα κράτη θα πρέπει να στηρίξουν τα μακροπρόθεσμα κοινωνικά κόστη. Όμως οι ασφαλιστές έχουν την σχετική γνώση. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει αυτή η σχέση έτσι ώστε η γνώση αυτή του ιδιωτικού τομέα να βοηθήσει τις κυβερνήσεις. Συχνά λέμε το ότι μόλις 10% πηγαίνει σε πρόληψη και 90% πηγαίνει στην αντιμετώπιση εκ των υστέρων των καταστροφών. Οι ασφαλιστές λοιπόν θα μπορούσαν να βοηθήσουν περισσότερο τα κράτη να αιτιολογήσουν ακριβώς το σκεπτικό του γιατί πρέπει να δοθούν περισσότερα χρήματα στην πρόληψη. Για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τώρα δεν θα αναφερθώ, απλά θα υπενθυμίσω ότι το 2007 είχαμε μια σχετικά νέα νέο κλάδο των ΑΠΕ και ε, αυτοί οι οποίοι την βοήθησαν τότε ήταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και είχε βοηθήσει πάρα πολύ στην τότε συγκυρία και είναι ακριβώς μεγάλος υπέρμαχος ε, της αύξησης του μεγέθους ε, τέτοιων επιχειρήσεων. Βεβαίως έχει και μεγάλο χαρτοφυλάκιο και τίθεται το ζήτημα και των άλλων δραστηριοτήτων της το θέμα τώρα της υποχρεωτικής ή μη αποκάλυψης. Δεν θέλω να πω ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο, αλλά ε, είναι η σχέση. Γιατί συχνά το εθελοντικό μας επιτρέπει να δούμε αυτό το οποίο θα μπορούσε να γίνει υποχρεωτικό. Και ο γαλλικός νόμος 173 είναι ένα παράδειγμα, όπου έχουν ένα παράδειγμα συμμόρφωσης ε, ή εξήγηση για την μη συμμόρφωση. Γιατί αν πάμε πάρα πολύ γρήγορα στο υποχρεωτικό μπορεί να είναι αναποτελεσματικό. Και έτσι θα δώσω τον λόγο στους ε, υπόλοιπους ε, μιλητές. Thank you very much, uh, so, Ο κύριος Αλιετά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ακούμε όμως ακόμα για ένα νέο κλάδο που πρέπει να αναπτυχθεί, εκείνον της πιστοποίησης. Γιατί το να δίνουμε κίνητρα εκπτώσεις ε, σημαίνει ότι συνεισφέρουμε στην κοινωνία, αλλά με έναν τρόπο απλώς που είναι αόρατος, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Δηλαδή δεν μπορούν να το λάβουν υπόψη τους απευθείας οι επιχειρήσεις. Αλλά εγώ αυτό που θέτω ως ιδέα ότι ακόμα περισσότερο από τη φορολόγηση του άνθρακα είναι να τοποθετήσουμε ένα στοιχείο άμεσης αποδοτικότητας για τους επενδυτές. Δηλαδή να έχουμε ένα κόστος της έκπτωσης του άνθρακα, ώστε να καθίσταται κίνητρο δηλαδή για τις επενδύσεις. Τα δυνητικά κενά που μπορούμε να έχουμε εκεί είναι ότι όλοι αυτοί που θέλουν να επενδύσουν στην ενεργειακή απόδοση είναι δώστε μου πιστώσει. Αλλά για να το αποφύγουμε αυτό πρέπει να έχουμε μια πιστοποίηση. Σχετικά δηλαδή με τον όγκο της πραγματικής μείωσης άνθρακα που έχει γίνει. Εάν θα μπορούσε λοιπόν να έχει ένα πιστοποιητικό μια επιχειρήση χωρίς να περιμένει την εισρωή ρευστού θα ήταν κάτι άμεσα πραγματοποιήσιμο για τους επενδυτές. Η πιστοποίηση λοιπόν θα πιστοποιούσε όγκους μείωσης εκπομπών διοξιδίου αερίων του θερμοκηπίου. Για την τράπεζα των επενδύσεων λοιπά Αυτό που μου φαίνεται πολύ σημαντικό στο σχέδιο Juncker είναι ότι πρέπει να έχουμε μια μεταρρύθμιση του σχεδίου. Δεν έχει κατεύθυνση. Είναι μόνο bottom-up αυτό το σχέδιο. Δηλαδή διαχειριζόμαστε τις επενδύσεις που εισραίουν. Αλλά δεν έχουμε μια, ένα σκεπτικό μιας βιομηχανικής πολιτικής πραγματικά. Μια κατεύθυνση, έναν άξονα. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει επενδύσεις από την αγορά οι οποίες θα μπορούσαν να περάσουν στο σχέδιο Juncker. Αλλά δεν υπάρχει μακροοικονομικό, με κριτήριο που να λέει θα κάνουμε μια βιομηχανική πολιτική, θα καλυφθήσουμε την τάδε κατεύθυνση. Δεύτερον, στοιχείο για να ενισχυθεί το σχέδιο αυτό. Πέρα από, τις, ε, από τα ε, πιστοτικά ιδρύματα, τα δημόσια, οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και ιδρύματα δεν συμμετέχουν στο στρατηγικό ταμείο επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν λάβουμε υπόψη μας όλες τις χώρες Έχουμε δημόσιες τράπεζες με παρελθόν πίσω τους. Εάν τους καταστήσουμε μετούχους του στρατηγικού ταμείου, τότε θα έχουμε ένα σημαντικό κεφάλαιο, αύξηση δηλαδή του κεφαλαίου της τράπεζας επενδύσεων και θα μπορούσε να έχει κανείς έναν όγκο κεφαλαίου δυνητικών επενδύσεων και να κατευθυνθούμε προς συγκεκριμένα έργα. και να πάμε στα 300, στα 500 και πιο ψηλά. Όμως, καθιστώντας τους μετόχους συνυπευθύνους άμεσα. Μια στρατηγική κατεύθυνση μια ενοποιημένη πολιτική. Υπό την ηγεσία και την κατεύθυνση τη Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριο Ράιν Κόλλεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να σα πω δύο λόγια για το θέμα των κρατικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε συνέχεια των όσων μα είπε ο Μισελ ε, βέβαια και συμφωνώ για το ότι η ΕΤΕ ε, θα πρέπει να επενδύει σε τομής ιδιωτική χρήσης του άντρακο. Το είπαμε και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι θέμα ευθύνης αυτών των ε, θεσμικών τραπεζών που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο κορβανά, οπότε υπάρχει αυτό το θέμα. Κατά πόσο δηλαδή, όπως λέει έκθεση, υπάρχουν αρκετά έργα να χρηματοδοτούν, γιατί είναι και θέμα ζήτηση, όχι μόνο προσφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Το οποίο σχετίζεται και βέβαια με τις πολιτικές λιτότητες τελευταία επτά ετία. Όμως τα κράτη έχουν την ευθύνη να δημιουργήσουν τις ευκαιρίες για ανανεώσιμες πηγές ενέργειες για μόνωση στα σπίτια. Στην Ελλάδα γενικότερα στο νότο της Ευρώπης Οπότε αν κανείς τάξει ένα τέτοιο στόχο, τότε κανείς έχει προσφορές από τον ειδικό τομέα. Οπότε η ΕΤΕ θα πάει προς χρηματοδότηση τέτοιων έργων. Βιώσιμο δηλαδή. Άρα έχουν σημαντικό ρόλο να διαμετρήσουν αυτές οι τράπεζες. Συμφωνώ με τον Μιζέλ. Δημιουργία δηλαδή δικτύου και στην κορυφή της πυραμίδας να είναι η ΕΚ. Τώρα στη συνέχεια του άλλου θέματος που αφορά αυτές τις κυρώσεις πράσινες, καφέ, τα είπε και ο πρόεδρος που μας είπε και τις προτιμήσεις του. Όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και έχουμε την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για αυτό το 25% δηλαδή είπαμε ότι τελικά ε, δεν έχουμε αποσπάσει τίποτα αποτελέσματα όσον αφορά την δανειοδότηση προς τις ΜΜΕ. 25, ούτε 50, ούτε 100. Επομένως, θα πρέπει να δούμε τι κεφάλαια μπορεί να υπάρχουν ως πράσινα δάνεια θεωρεί και ο κόσμος ότι έχουν απαραίτητη κεφαλαιοποίηση οι τράπεζες. Δηλαδή, ναι, να πάνε επιστώσει στον πράσινο τομέα, αλλά να υπάρχει και η ζήτηση. Αλλιώς, αυτή η προσέγγιση είναι ρηψοκίνδυνη και επομένω είναι win-win η επιβολή των καφέ κυρώσεων. τέτοιο καφέ στοιχεία ενεργητικού. Να πάμε σε περισσότερη ευελιξία και θα πρέπει ίσως να αναθεωρηθούν γενικότερα και οι πολιτικές δανειοδότηση. Κύριο Φέρμπερ που πρόεδρε, ευχαριστούμε που ήρθατε στην ακρόασή μας, συνεχίζουμε τώρα με το θέμα, αλλά τώρα επί τη βάση μιας έκθεσης, της έκθεσης της κυρίας Μόλι Σκοτ Κέιτον. Και πάλι ευχαριστούμε που ήρθατε. Perhaps ask if we might be back in touch with you if we could use your help in future. Thank you. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και επιφυλασσόμεθα να πείθουμε σας και στο μέλλον. Πολύ συναρπαστική καιρή που ζούμε όσον αφορά το ότι τώρα χρειάζεται να γίνει κάτι για το κλίμα μετά από δεκαετίες να δούμε από λεβάς βιομηχανίας, μείωση των εκπομπών από διάφορες βιομηχανίες, βιομηχανίας, να δούμε τι μπορεί να γίνει όσον αφορά την χρηματοδότηση, είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, ούτως ώστε να επιταχύνουμε την μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον και η Συμφωνία των Παρισιών έχει δώσει καινούργια όθηση σε αυτή την υπόθεση. Άρα θα πρέπει το Κοινοβούλιο να διαμορφώσει μια κοινή θέση. Πώς το χρηματοοικονομικό σύστημα να βοηθήσει και να μην εφραγμόσει αυτή την μετάβαση. Όπως ήδη είπαν οι προσκεκλημένοι μας, θα πρέπει με τα όσα έχουν ε, συμμετεί για το κλίμα να είναι συμβατές οι πολιτικές δανειοδότησες. Όπως επίσης και τα κριτήρια της εταιρική διακυβέρνησης, άρα να έχουμε κάποιους στόχους που να οδηγούν σε ε, επενδύσεις 4,7 έως 6,7 3 ε, εκατομμύριων για να μπορούμε να πάμε στους βιώσιμού, στο Άρα και η βιώσιμη χρηματοδότηση θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο και έτσι τα κεφάλαια να πηγαίνουν προς τις αναγκαίες επενδύσεις για μια ταχεία δίκαιη μετάβαση την οικονομία και για την κοινωνία. Οπότε η Ευρώπη να έχει πάλι πρωτοπορία για την αλλαγή του κλίματος και έτσι να είναι ακαίρεση οι αξίες μας και επίσης το πλεονέκτημα της βιομηχανία μας. Επομένως, συμφωνούμε με τόσο είπε η ομάδα υψηλού επίπεδου. Στην έκθεση λέμε ότι προσβλέπουν στα θεσμικά όργανα της Ένωσης οι πολίτες της Ένωσης. Θέλουμε τα χρήματα που υπάρχουν να οδηγήσουν σε σταθερό κλίμα και προστασία του οικοσυστήματος που θα ωφελήσει σημερινές και τις μέλουσες γενναίες. Τώρα μέχρι να με κόψει ο πρόεδρος θα σας πω τα Πρώτον, θα πρέπει να δούμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει αποκάλυψη όσον αφορά κάποια δεσμευμένα στοιχεία του ενεργητικού σε σχέση με την οδηγία για λογιστική και χρηματοοικονομικά. Όσο αποφάσισαν οι G20 να συνεχιστούν οι υποχρεώσεις ε, των καταπιστευματοδόχων και να υπάρχουν πληροφορίες για πάσα προσφορά για κάθε επένδυση. Όλοι να μπορούν να έχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την ταξόνομη. Ακούσαμε τι προσφέρουν πολιτικές ομάδες και θέλουμε να καθοριστούν κάποια κριτήρια, κάποιους μεταβλητές, να γίνει η κατάσταση πιο δυναμική, να αξιοποιηθεί παν στοιχείο ενεργειακού. Συνταξιοδοτικά, επενδυτικά προϊόντα να ληφθούν υπόψη, αλλά προσοχή, προσοχή όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια και τα ορυκτά καύσιμα μείνουν απ' έξω. Επομένω, σε αυτό το δυναμικό πλαίσιο πιο σωστά είναι να έχουμε διαφορετικά πρότυπα, τρία. Το ελάχιστο, σύμφωνα με το όσο είπαμε στο Παρίσι, σύμφωνα με την ανάλυση ESG και σαν ενδιάμεσο να έχουμε κάποιες δραστηριότητε που οδηγούν σε επιπτώσεις θετικές όπως πρωτοβουλία για τη χρηματοδότηση αλλά επίσης να καλύψουμε δραστηριότητες που θα οδηγούν σε μια θετική μετάβαση και οικολογική αναγέννηση. Να εξασφαλίσουμε επίσης ότι είναι παραδείγμα προς μίμηση τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, κυρίως η ΕΤΕ και η κάπατα. Να καλύπτουν τα κενά των άλλων και ό,τι να υπάρχουν για τις δεσμεύσεις τους. Επομένως, και οι στόχοι ESG θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις δεσμεύσεις του Παρισιού στο μέλλον. Να έχουμε δανεισμό μόνο συμβατό με τη Συμφωνία των Παρισίων. Προς νομοκρατικές τράπεζες και η πενετική πολιτική να είναι συμβατή με αυτούς τους στόχους ESG. Ευχαριστώ και πάλι τους και οδησίγητες σίγουρα μπορούμε να διαμορφώσουμε μια ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου και έτσι να μπορούμε από θέση ισχύω τον Μάιο να μιλήσουμε στην Κομισιόν, να τάξουμε επομένω τους στόχους που πρέπει και έτσι με την Κομισιόν, μόλι κατεβάσει την πρότασή τη να έχουμε έναν παραγωγικό θετικό διάλογο. Ο Πρόεδρος. Ποιητικά η κυρία τι κάνει. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κοιτώντας ε, και το ρολόι θα αφήσω τα γενικά σχόλια και τα συγχαρητήρια για την ε, εργασία της εισηγήτριας και κάποια γενικότερα θέματα. Θα ξεκινήσω με τους ε, δείκτες. Δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που θα κάνω τέτοια μνήα. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε πραγματικά να ενσωματώσουμε την ιδέα των δικτών ως αρχή κριτήριο λογιστικής, ε, λογιστικού ελέγχου. Όσο ασχολούμαστε μόνο με την ορολογία και την ονοματοθεσία αφήνουμε τον κλάδο ελεύθερο. Ούτως ή άλλως θα, υπάρχει, θα εξακολουθήσει να υπάρχει κατασκευαστική διαδικασία και χρήση του μπετόν, για να το πούμε έτσι. Όμως αν δεν συγκρίνουμε τις επιχειρήσεις, τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές μεταξύ τους, δεν πρόκειται να έχουμε πραγματική μεταμόρφωση της ε, βιομηχανίας του κλάδου αν απλώς υιοθετήσουμε μια ορολογία, μια ονοματολογία. Δηλαδή ότι δίνουμε μια ετικέτα σε κάτι ότι είναι πράσινο. αυτός ο παράγοντας στήριξης, ο πράσινος παράγοντας στήριξης και αυτό ε, εγείρει ερωτηματικά γιατί κανονικά δεν πρέπει να αναμειγνύουμε τους δείκτες οικονομικής επίδοσης και πράσινης ή περιβαλλοντικής επίδοσης. Γιατί μάλλον το να θέτουμε κεφαλαϊκά κριτήρια τελείως διαφορετικά είναι εσφαλμένο και αυτό ε, αφορά και στην ε, λειτουργία της ίδιας της ε, Κεντρικής Τράπεζας. Αν γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια εναλλακτική εγγύηση που θα αγοραστεί από την <coughs> ΕΚΤ οποιασδήποτε ετικέτας πράσινης, τότε είναι αντικίνητρο. Αυτές είναι κάποιες από τις βασικές μου ανησυχίες, συν το εξής. θα πρέπει να αφήσουμε επαρκή ευελιξία για το μέλλον και τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις να βρουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μάλιστα ιδιαίτερα σκεπτόμενοι τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους ε, μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων. Άρα το comply or explain και όχι το comply μόνο του θα έπρεπε εκεί να υπερισχύει. Για τον ε, ρόλο και τη λειτουργία των ασφαλίσεων η κάλυψη κάθε περιβαλλοντικής ευθύνη είναι ένα στοιχείο που θα έπρεπε να εξετάζουμε και να μην ξεκινούμε και να τελειώνουμε με το διοξείδιο του άνθρακα διότι υπάρχουν δραστηριότητες ε, ε, στην οικονομία της βιοπικιλότητας που δεν πρέπει να τους περιορίζουμε για να μην δημιουργήσουμε άλλη μια κατηγορία δηλαδή ε, παγωμένων σταθερών περιουσιακών στοιχείων. Ε, συνολικά πάντως είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η δουλειά και πνευματικά πραγματική πρόκληση, αλλά περιμένω με ενδιαφέρον και την συζήτηση των υπολείπων ε, εισηγητών και τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ο κύριος Στάγνη. Ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή έκθεση. Έχουμε μια ένα πολύ καλό κείμενο της Μόλις Σκότ και πρέπει να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να φτάσουμε σε μια πλήρη αλλά και ευέλικτη προσέγγιση ώστε να αλλάξουμε τον κόσμο των χρηματοπιστωτικών ε, και να του ορίσουμε μια κατεύθυνση. Είναι μια δύσκολη και περίπλοκη δουλειά και έχουμε ήδη καθυστερήσει αλλά καλό είναι να την κάνουμε. Γιατί πρέπει. Και αυτό απαιτεί αλλαγές για πάρα πολλά επίπεδα συμμετοχής στα χρηματοπιστωτικά. Τράπεζες, ασφαλιστές, διαχειριστές ε, περιουσιακών στοιχείων, ε, ο, οίκους αξιολόγησης, ε, αρχές ε, επιμέλειας και επιτήρησης. Όλοι αυτοί θα πρέπει από κοινού να εξασφαλίσουν ότι δεν θα είναι ένα, απλώς ένα θέμα καλής θέλησης αλλά ότι θα μεταφράζεται σε αυτά μέτρα σε πραγματικότητα δηλαδή. Και νομίζω ότι και η Κεντρική Τράπεζα έχει κεντρικό ρόλο να διαδραματίσει εδώ, ώστε να συλλέξει αυτές τις βέλτιστες πρακτικές για να τις υλοποιήσει. Τώρα εξετάζω και εγώ τρόπους το σύστημα να μην είναι εθελοντικό. Να είναι, να έχει περισσότερα στοιχεία δεσμευτικότητας. Ίσως τα κίνητρα θα πρέπει να είναι περισσότερα το νομοσχέδιο 173 το γαλλικό είναι ενδιαφέρον αλλά ίσως το διοικητικό συμβούλιο και οι ενδιαφέροντες σύμβουλοι πρέπει να καθίστανται υπεύθυνοι Δηλαδή ζητούμε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από τους μετόχους, λέει ο μιλτής, να κατανοήσουν τους κινδύνους αυτούς και να τους ενσωματώσουν στις αποφάσεις τους. Και πρέπει να κοιτούμε και τα πακέτα αμοιβών. Ε, για να μην δίνουμε αντικίνητρα Για να μην έχουμε δηλαδή αντίκτυπο επί της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού κλάδου και πάλι εκτός από το περιβάλλον. Και το τελευταίο μου σχόλιο, νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να δώσουν ένα παράδειγμα οι χρηματοπιστωτικοί φορείς θα πρέπει να υλοποιήσουν τις βελτιστές πρακτικές αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι και η Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πρότυπα. Θα έπρεπε να είναι πρότυπα και θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι φορείς που θα εφάρμοζαν τα συμπεφωνημένα αυτά κριτήρια. θα μπορούσαν πράγματι να έχουν σημαντικό αντίκτυπο δείχνοντας την κατεύθυνση στον κλάδο. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί κανείς να το τονίσει επαρκώς. Ευχαριστώ. Uh, uh, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για την συζήτηση αυτή, την επικοδομητική. Ωραία. Θα προλάβουμε κιόλας. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σας κυρία Σκότ για το σχέδιο έκθεσης. Αντικατοπτρίζει τους κοινού μας ε, στόχους. Ε, πρώτα απ' όλα δηλαδή να ενισχύσουμε την σταθερότητα και την βιωσιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και δεύτερον να κατευθύνουμε περισσότερα κονδύλια προς τις βιώσιμε επενδύσει. Θεωρώ ότι η στόχη αυτή είναι συμπληρωματική. Πώς θα τους πετύχουμε όμως. Είναι αφελέ να θεωρούμε ότι οι περισσότεροι επενδυτέ θα επενδύσουν σε βιώσιμα προϊόντα χάρη της ε, αηφορία. Δεν θα το κάνουν και δεν θα έπρεπε να το κάνουν. Θα έπρεπε να επενδύουν σε αυτά γιατί είναι πιο επικερδή και λιγότερο επικίνδυνα. Ως ε, νομοθέτες είναι η δουλειά μας να διασφαλίσουμε ότι θα συμβαίνει αυτό κατά το οποίο συμβαίνει μέσω διαφόρων νομοθετημάτων όπω το σύστημα ETS. Ε Επίσης η έκθεση αυτή δεν είναι το σημείο στο οποίο θα ορίσουμε άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Τι μπορούμε να κάνουμε. Θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα την πραγματική του τιμή και οι επενδυτές να έχουν επαρκείς πληροφορίες από τον κλάδο ε, υπάρχει μια υποχρέωση να λάβουν υπόψη του σχετικούς παραγόντες όπου αυτό ισχύει και μια κατηγοριοποίηση που θα τους υποχρεώνει να συγκρίνουν και να καθορίζουν τα διαφορετικά προϊόντα επιπλέον. Όταν έχουμε ένα σύστημα κατηγοριοποίησης λέτε ότι χρειαζόμαστε ένα ευέλικτο πλαίσιο συμφωνώ αλλά συνειδητοποιώ επίσης ότι αυτό θα απαιτήσει ένα σύστημα διακυβέρνησης. Έχετε μια πρόταση, μια ιδέα για το τι μορφή θα έχει αυτό. θα ήταν δημόσια, ιδιωτική πρωτοβουλία ή μια σύμπραξη και πώς θα διασφαλίσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους ενδιαφερόμενους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σοβαρεμούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο την Σκότια για τον ε, φάκελο που έχει ετοιμάσει ως οικειώδης εισηγητής. Ε, να πω ότι Κατά την άποψή μου η δουλειά που έχει κάνει κινείται σε μια θετική κατεύθυνση ε, και σκοπεύω και στην φάση των τροπολογιών να συμβάλλω επικοδομητικά ε, έτσι ώστε στο τέλος με την ευρύτερη δυνατή συνένεση να εγκρίνουμε μια καλή έκθεση. Ακούγοντας ορισμένους από τους σκιώδεις συγητές ορισμένων πολιτικών ομάδων μου δημιουργήθηκε το ερώτημα αν πραγματικά πιστεύουν στη Συμφωνία του Παρισιού. Εάν πραγματικά αυτό που είναι η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμβατότητά της με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού αλλά και με τους αναπτυξιακούς στόχους του ΟΗΕ μας απασχολεί όλους πώς, θα το πετύχουμε. Έχω διαβάσει πάρα πολλές απόψεις οικονομολόγων που λένε ότι επενδύοντας στην πράσινη ανάπτυξη μπορούμε να έχουμε και κέρδη και απασχόληση. Αλλά χρειάζεται να δούμε και τα εργαλεία που θα βοηθήσουν τον αναπροσανατολισμό των επενδύσεων. Ακούσαμε προηγουμένως εισηγητές στο hearing που ήταν για το ίδιο θέμα, που με τεκμηρίωση μας είπαν αυτά τα πράγματα. Αν μείνουμε απλώς σε μία νοοτροπία υπερφιλελεύθερη, όπου απολυτοποιούμε μόνο το κέρδος και δεν μας ενδιαφέρει το περιβάλλον, η δημόσια υγεία, η επένδυση στην καινοτομία προκειμένου να δημιουργήσουμε συμβατές με την προστασία του περιβάλλοντος μορφές οικονομικής ανάπτυξης, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Τότε επιβαρύνουμε το περιβάλλον, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τη δημόσια υγεία και αφήνουμε άλλες χώρες, οι δυνάμεις περιφερειακές, ανταγωνιστικές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κερδίζουν έδαφος στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται να βρούμε εργαλεία, δείκτες βιωσιμότητας, σχήματα που να υπηρετήσουν τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προσυπογράφοντας τη Συμφωνία του Παρισιού. Που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνώντας με τους αναπτυξιακούς στόχους του ΟΗΕ. Και σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο, από ό,τι θυμάμαι, και παλιότερα που ήμουν μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, είχε ένα ρόλο πρωτοπορίας. Πίεζε την Κομισιόν και το Συμβούλιο να κάνουν πράγματα. Και όχι ένα ρόλο φρένου, ένα ρόλο ανάσχεσης. Θα ήθελα λοιπόν από όλους μας να καταθέσουμε και προτάσεις και εκτός από ερωτήματα δυσπιστίας ή άρνησης να, να καταθέσει ο καθένας προτάσεις επικοδομητικές προς την έκθεση της κυρίας Σκοτ για το πώς μπορούν να υπηρετηθούν αυτοί οι στόχοι με τρόπους συμβατούς με τη φιλοσοφία και το πολιτικό πρόγραμμα της πολιτικής του ομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Και περνάμε τώρα στο KHDI. Ο Σβεν Γκίγκολντ είναι στη λίστα μου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και επίση να μην παρατηρήσεις θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι η πολιτική ατμόσφαιρα άλλαξε τα τελευταία χρόνια όσον αφορά αυτή την πρόταση. Πριν από λίγα χρόνια η χρηματοδότηση, η πράσινη, ήταν κάτι το μη απαραίτητο, κάτι το μυστηριώδες. Να τώρα βλέπουμε όμως πως όλοι ποθούν για κάτι τέτοιο ή, ε, όσον αφορά τη ζήτηση και όσον αφορά την προσφορά χρηματοοικονομικών προϊόντων. Άρα χρειάζονται στεχνοί κανόνες από την Ένωση και αυτοί οι κανόνες θα κάνουν τη διαφορά. Ήδη διεθνώς ε, έχουμε ε, για τα UCIT ένα πλαίσιο ε, και έτσι μπορεί να έχουμε πράσινα προϊόντα και να πετύχει το εγχείρημα αυτό εάν είναι εύστοχοι οι κανόνες που θεσπίσουμε. Επίσης και συμφωνώ με αυτά που είπε ο συναδελφός της Άλντε ότι η πράσινη χρηματοδότηση ποτέ δεν θα αντικαταστήσει την οικολογική πολιτική, την οικολογική κατανάλωση και παραγωγή Θέλουμε κάποιες επιλογές που να είναι κερδοφόρες. Ε, άρα και τα προϊόντα, τα οικονομικά να μπορούν να επιστρατευτούν. Και άλλο αυτό και άλλο η χρηματοδότηση. Άρα να έχουμε ένα νομικό πλαίσιο, διάφανο, ξεκάθαρα ε, πρότυπα, ούτω ώστε να κάνουμε αυτά που είπε ο Πολ, τάν για τους ε, κινδύνους Άλλο αυτό όμως και άλλο οι κεφαλαιακές απαιτήσει, όπως είπε ο συνάδελφος από το ΕΛΚ. Πράσινη οικονομία σημαίνει καινοτομία. Υπάρχουν όμως κίνδυνοι εδώ, ίσως υπάρχουν ακόμη περισσότεροι κίνδυνοι από ότι ε, στις άλλες επιλογές. Οπότε γι' αυτό και κάθισα και άκουσα τι είπε ο πρόεδρος μας ε, στα μέσα ενημέρωσης. Το είπε και ο Μαρκούς Φέρμπερ. Και άλλο κεφαλιακές απαιτήσει και άλλο πράσινα προϊόντα χρηματοοικονομικά. Σε άκουσα, σε άκουσα, Μάρκος. Πρέπει αυτά να τα ξεχωρίζουμε. Άλλο η οικολογία και άλλο το πώς θα ρυθμίσουμε τα των ασφαλιών, τα των τραπεζών κλπ. Προσοχή επομένως κεφαλιακές απαιτήσει να μην είναι κάποιο είδου ε, ευκαιρία και κάτι δούριο ύπος για κάθε είδου ε, επιχειρηματία. Άρα, προσοχή, όπως είπε ο Πολτάνκ, και να κάνουμε αυτή την ε, διάκριση. Στον αφορά τις κεφαλικές απαιτήσεις. Ο πρόεδρος, α, τώρα, τώρα κατάλαβα. Κατάλαβα τι είπα. Έχουμε εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ο Πρόεδρος. Θέλετε να μας μιλήσετε. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Welcome very much. Θα είμαι σύντομο. Ε, χαιρετίζουμε την έκθεση της ε, εισηγητρία και εργαζόμαστε σκληρά για να κάνουμε και το σχετικό follow-up της έκθεσης της ομάδας υψηλού επίπεδου ώστε να έχουμε ένα σχέδιο για τη βιώσιμη χρηματοδότηση εντός του πρώτου δεκαπενθημέρι του Μαρτίου. Αυτό το έγγραφο λοιπόν θα θέσει το πλαίσιο και για τη βιώσιμη χρηματοδότηση ευρύτερα και διεθνώς. Θα διοργανωθεί και ένα συνέδριο υψηλού 22 Μαρτίου και θα έχουμε τέσσερις προσκεκλημένους υψηλότητα του επίπεδο από το Κοινοβούλιο και περιμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχιση της συνεργασίας μας. Σας ευχαριστώ. Ξαναδίνω τώρα το λόγο στην Μόλη. Ευχαριστώ Μάκους. Είναι πράγματι σπάνιο σε τόσο αντιφατικό ζήτημα να υπάρχει τόσο καλή βούληση και συμφωνία αλλά θα θέσω και ένα-δύο θεματάκια που θα διασκεδάσουμε και με τους σκιώδεις μετά. Καταρχάς έχουμε αυτό το θέμα της, ε, της ε, κατάταξης. Ε, αυτό το θέμα των δικτών είναι σημαντικό. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να μετακινήσετε το 80% στο μέσον και να μην ανησυχείτε για τα δύο άκρα, αλλά πρέπει να μπορούμε να έχουμε μια ετικέτα, μια επισήμανση πρέπει να μπορούμε να λέμε ότι εμείς πιστοποιούμε το χ προϊόν ως πράσινο, γιατί η αγορά δεν έχει καταφέρει να πείσει τους επενδυτές για το τι είναι πράσινη επένδυση. Αν δεν έχουμε λοιπόν ένα αξιόπιστο σήμα, τότε οι Κινέζοι εκδίδουν διάφορα ομόλογα πράσινη επένδυση που στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου πράσινη. Επομένω, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ορίζουμε κάτι ένα σήμα, μια πιστοποίηση με την ευρωπαϊκή αξιοπιστία πίσω του ως πράσινο. Τώρα έγινε μια ερώτηση για το ποιος θα το διοργανώσει αυτό. Έχουμε εμπειρογνώμονες και ε, διοργανώνουμε μια ομάδα με προσκεκλημένους ενδιαφερόμενους φορείς. Αυτό είναι ανοιχτό ζήτημα, αλλά πρέπει να βασιστούμε καταρχάς στις επιστημονικές ενδείξεις για το τι είναι ασφαλής και μακροχρόνια και βιώσιμη επένδυση και τι δεν είναι. Τώρα για τον παράγοντα πράσινο κάθετος καφέ. Έχουμε και τη μελέτη του LSE που δείχνει ότι χρειάζεται να καταβληθούν τεράστιες προσπάθειες ώστε να μειώνονται οι κεφαλαϊκές απαιτήσει σχετικά με τις πράσινες εμερνήσεις και πρέπει να συμφωνήσω με τον Σβέν, δηλαδή συμφωνώ μαζί του, ότι εδώ ανοίγουμε ένα επικίνδυνο παράθυρο. Ότι δηλαδή εφόσον εγκρίνεται όσα κάνουμε θα βλέπουμε και εμείς πιο επίοικο στις κεφαλαϊκές απαιτήσει. Δεν θα έχουμε δηλαδή ε, ανασταθεροποιήσει με επαρκώς αξιόπιστο τρόπο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στην, στην πραγματικότητα σήμερα δεν συνυπολογίζουμε το κόστος της υπεύθυνη και βιώσιμης ε, ε, πράσινης επένδυσης σήμερα. Υπάρχουν τεράστιοι κίνδυνοι στο σύστημα με διάφορα κατακαιρματισμένα περιουσιακά στοιχεία. Μέχρι στιγμής έχουμε επικεντρωθεί στα θέματα του άνθρακα, αλλά έχουμε διαχείριση γεών, εδαφών, αλληλείας κτλ. Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι δεν έχουν αποτυπωθεί με ακρίβεια, με επάρκεια. Πρέπει λοιπόν να γίνει αυτό, να υπολογιστούν αυτοί οι συστημικοί κίνδυνοι της ζωής στον πλανήτη και κατά τα άλλα ευχαριστώ όλους για τα καλά τους λόγια και την ε, συνέχιση της συνεργασίας μας ε, και στις ε, συναντήσεις των σχεδόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ Μόλι. Λέει ο Πρόεδρος, ήσασταν τόσο αποτελεσματικοί που είμαστε στο χρονοδιάγραμμα. Τόσο καλοί είμαστε που δεν έχουν φτάσει οι επόμενοι ομιλητές. Τέλος πάντων, για τις ε, τροπολογίες 31 ε, Μαρτίου 12 το μεσημέρι και ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ τέλη Απριλίου και 26 Μαρτίου η εξέταση τροπολογιών. Επομένως, έχετε χρόνο να υποβάλλετε τροπολογίες για τη μόλη. Το επόμενο σημείο είναι η συζήτηση για την ε, μόνιμη θέση στο ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης. Ε, θα κάνουμε μια, ένα σύντομο διάλειμμα ίσως, ελπίζοντας ότι οι συνάδελφοι που έχουν οριστεί να συζητήσουν το θέμα αυτό θα προσέλθουν.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 Uh, Συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Δεν χάνουμε καθόλου καιρό. Περνάμε σημείο 13 και τυχερό έχουμε προτινόμενο υποψήφιο για θέση στο Δέλτα Σίγμα του Συμβουλίου Διάσωσης ε, Τραπεζών. Καλωσορίζουμε ορίζουμε τον υποψήφιο της του Συμβουλίου ε, Έχουμε τον υποψήφιο της Κομισιόν, ο κ. Γιάννη Γιάννης Πεκ, ο οποίος είναι διοικητής της Τράπεζας της Σλοβενίας. Καλώς ήρθατε λοιπόν. και ήδη τα άλλα μέλη της Ομάδας Εργασίας Τραπεζικής Ένωσης είχαν στις 21 Ιανουαρίου μια συνάντηση και κλεισμένων των θυρών. Η δεύτερη φάση της επίσημης επρόασης είναι τώρα δημόσια και είχε ένα σημαντικό ρόλο καθώς τονίζει την λογοδοσία των μελών του ενιαίου αυτού Συμβουλίου Και βεβαίως η εκρόση έχει μεγάλη σημασία για το αν θα εγκρίνουμε τον υποψήφιο της Κομισιόν καθώς μετά θα ψηφίσουμε. Προτείνω λοιπόν να ξεκινήσετε εσείς και μετά να έχουμε ερωτήσεις ε, με τη γνωστή διαδικασία 5 λεπτά για ερώτηση και απάντηση οπότε όσο πιο πολύ ρωτάτε τόσο πιο σύντομη θα είναι η απάντηση απλό και με χαρά τώρα σας δίνω τον λόγο κύριε Γιάσπετς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Μπούστον Γιάσπετς λέγονται, λέγομαι, διοικητής της ε, Τράπεζας της ε, Σλοβενίας, μέλος του Δουσού της ΕΚΤΟ. όπως έχω πει πολλές φορές, ξεκίνησα την ζωή μου ενήλικος ε, πεπισμένος ότι θα γίνω μουσικός όμως μια νύχτα έγινα οικονομολόγος και κεντρικός τραπεζίτης, κάτι το οποίο δεν έχω μετανιώσει ακόμα και θεωρώ πως ε, αυτό το οποίο έκανα στην σταδιοδρομία μου με καθιστά ικανό να καταλάβω αυτήν την θέση. Μετά τις σπουδές μου λοιπόν έκανα για λίγο καιρό έρευνα πανεπιστημιακή και μετά ενταχθήκα στην ε, τράπεζα της ε, Σλοβενίας σε νεαρή ηλικία έχοντας την ευκαιρία και το προνόμιο να συνεργαστώ με τους ε, συναδέλφους μου, τους συμπατριώτες μου σε μια εποχή στην οποία έμπαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Σλοβενία και ήταν η πρώτη χώρα που υιοθέτησε το ευρώ το 2007. Το 2009 πήγα στο Δελτανιτάφος σύμβουλος ε, της ε, Κεντρικής Τράπεζας του Κοσφοπεδίου για τέσσερα χρόνια και μετά εργάστηκα ως ε, σύμβουλος στην Κεντρική Τράπεζα του Σουρινάμ και τέλος έγινα τον Ιούλιο του 2013 διοικητής της Τράπεζας της Σλοβενίας το μέσο κρίσης όταν η Σλοβενία θεωρείται άλλη μια χώρα στο σε πρόγραμμα και επιτυχώς με την κυβέρνηση παλέψαμε και κυριολεκτικά σώσαμε την χώρα. Και έτσι σήμερα έχουμε θα έλεγα ένα χαρακτηριστικό υπόδειγμα του πώς η αργή αντίδραση μπορεί να κοστίζει περισσότερο και το πώς βεβαίως ναι, μια χώρα μπορεί να τα πάει μετά καλύτερα. Βεβαίω δεν συμφωνούν όλοι με τα όσα κάναμε στην ε, Σλοβενία. Ε, ειδικά το Μπέιλιν, αλλά συμφωνούμε με το πλαίσιο το οποίο έχουμε σήμερα, τους ίσους όρους ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη και νομίζω ότι στόχο έχει να προστατεύσει ακριβώς τους ε, φορολογούμενους και να διασφαλίσει την η οικονομική σταθερότητα της χώρας και της Ευρωζώνης γενικότερα. Θα σταματήσω τώρα εδώ και είμαι στην διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε κύριε Γιάσμπετς. Και τώρα, για το... ο κύριος Μπάλτς για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ε, καλώς ήρθατε. Θα ήθελα να αναφέρω κάποιες σκέψεις μου για το καθεστώς αυτό της αναδιάρθρωσης και να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας. Θεωρώ ότι είναι σαφές ότι, ένα, ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο αποτελεσματικό καθεστώς ε, με απλούς ε, κανόνες ε, και κυρίως να μειώνει τους κινδύνους για μια δύσκολη διάσωση ή και χρεοκοπία τραπεζών. Δεν θα πρέπει όμως να πέσουμε κάτω από την παρδιαγραφή MRL της BRD, αλλά θα πρέπει αυτό να αποτελέσει την αφετηρία μας για περαιτέρω ενίσχυση των διατάξεων του Άμπρελ. Και θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι όσον αφορά την ποιότητα του Άμπρελ, παραδείγματος χάρη. Εδώ πέρα κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές για την κατάταξη έχουν μεγάλη σημασία και θα πρέπει να περιορίσουμε εκ των προτέρων την ποιότητα. Μετά. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να έχουμε ένα στο δυνατόν ευρύτερο moratorium για να ενισχύσουμε την δυνατότητα παραμβάσεων και να μην περιορίσουμε εκ των προτέρων. Αυτές ήταν οι σκέψεις μου. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Τι ε, τοποθέτηση έχετε εσείς ε, ως προς αυτά και ε, τι θεωρείτε ότι θα χρειαζόμασταν επιπλέον. Ευχαριστώ. Uh, uh, uh, Ευχαριστώ τον κύριο Μπάλς. Ε, νομίζω ότι θέτεται ένα σημαντικό ερώτημα. Καταρχά ε, για τον μηχανισμό εξυγένσης. Όπως έχει σήμερα στο χαρτί, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε. Το ζητούμενο είναι η υλοποίηση και το ακόμα μη λυμένο πρόβλημα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες δικαιοδοσίες που δεν συμμετέχουν πλήρως στο παρόν σύστημα επίλυσης διαφορών. Χρειαζόμαστε <clears throat> περισσότερη συνεργασία μεταξύ, για να το θέσω έτσι και επιτρέψτε μου, Φραγκφούρτης και Βρυξελών. Μεταξύ Κεντρικής Τράπεζας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με όλους τους δορυφορικούς οργανισμούς τους, που ένας από αυτούς είναι και το ενίο Συμβούλιο Εξηγένσης. <clears throat> Νομίζω ότι πλησιάζουμε προς μια τέτοια κατεύθυνση, αργά αλλά σταθερά, έχουμε και διδάγματα και εμπειρίες από το παρελθόν και νομίζω ότι υπό την έννοια αυτή αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να υλοποιήσουμε τις δυνατότητες <clears throat> επίλυσης διαφορών που έχουμε στην νομοθεσία. Και νομίζω ότι επ' αυτού ελπίζω να απάντησα δηλαδή. Για το MREL είναι ένα ευαίσθητο θέμα αλλά η εισαγωγή του θα μπορούσε να επιφέρει χρηματοπιστωτική αστάθεια και όχι σταθερότητα αν δεν είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχουν κάποια τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες, των οποίων οι τράπεζες δεν είναι σε θέση να συμμορφωθούν πλήρως με το σημερινό καθεστώς ΕΜΡΕΛ. και το να τις εξωθήσουμε θα μπορούσε να τις οδηγήσει σε αστάθεια. Βεβαίως από την άλλη μεριά το Έμρελ είναι εκεί και θα παραμείνει εκεί, είναι απλά ζήτημα του πότε θα μπορέσουμε να, το, να ενσωματώσουμε και κάποιες άλλες δικαιοδοσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό. Για το τρίτο ζήτημα, το moratorium, γνωρίζετε πώς υπολογίζεται αυτό σε διάφορες χώρες. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Δίνει χρόνο επαρκούς και ενδελεχούς εξέταση δεδομένων και δίνει και στους ηθήνοντες σε αυτή την περίπτωση SSM και SRB επαρκή χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουν και να οργανώσουν καλύτερα τα συχνά οδυνηρά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Υπάρχει όμως ελπίδα να κινηθούμε σε μια σωστή κατεύθυνση. Λοιπόν, είχαμε αυτά τα πεντά λεπτά για να μην τα υπερβαίνουμε πάρα πολύ. Ο κύριος φων και έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλωσορίζω τον υποψήφιο. Έχω τρεις ερωτήσεις. Καταρχάς μία ε, ερώτηση που απορρέει από την παρατήρηση του κυρίου Μπάλτς για το MRL. Έχουμε μία επιλογή στην υφιστάμενη νομοθεσία μας. Πόσο αυστηροί θα είμαστε, πόσο εξαντλητικοί θα είμαστε επί του Έμρελ. Τώρα, αν κάνουμε ταχαίω πράγματα που είναι δύσκολα για τράπεζες που δεν είναι απολύτως υγιείς, ναι, αυτό θα ήταν πρόβλημα. Από την άλλη, αν αφήσουμε πολύ μεγάλο ε, περιθώριο ευχέρειας, τότε δεν κάνουμε επαρκή πράγματα υπό την έννοια της εξυγέννησης. Και επομένως Πού βλέπετε αυτή τη γραμμή ισορροπίας, γιατί αυτό πρέπει να διατηρούν υπόψη οι νομοθέτες. Και αυτό θα είναι και ένα από τα βασικά σας προβλήματα αν αποκτήσετε αυτή τη θέση που φιλοδοξείτε. Σε πιο πρακτικό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια είχαμε ήδη μια κάποια εμπειρία με το νέο καθεστώς με την Τραπεζική Ένωση με την Banco Popular, με κάποιες, μια δύο στην Ιταλία και διαρωτώ με εσείς από αυτές τις εμπειρίες τι θεωρείτε ότι μπορούμε να αντλήσουμε ως δίδαγμα για το μέλλον. Και κάτι για το οποίο εγώ προσωπικά ανησυχώ. Εσείς τι θεωρείτε, ποια θεωρείτε ότι θα είναι η επίπτωση του Brexit επί του πλαισίου εξυγίανσης. Ευχαριστώ κύριε Φων Βάιστσεκα για τα ερωτήματα αυτά, τα τρία αυτά ερωτήματα. Ε, θα απαντήσω χωρίς βέβαια να δίνω τελεσίδικες ή απόλυτα πλήρες απαντήσεις αυτή τη στιγμή. Για το Έμρελ να σας πω το εξής έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε το διαρκές δίλημα αυστηρότητα έναντι περιθωρίου. Η μόνη διέξοδος είναι η καλύτερη διαχείριση του χρονικού ορίου εντός του οποίου θα πρέπει να συμμορφωθούν πλήρως με το έμρελ. Είναι βεβαίως δύσκολο, ιδιαίτερα σεβόμενος κανείς ισότιμους κανόνες παιχνιδιού για όλους, αλλά σε κάποιες χώρες όπως είπα, κατά την άποψή μου, το να ε, εξωθήσουμε πλήρως σε πλήρη συμμόρφωση και εισαγωγή του Έμρελ θα μπορούσε να οδηγήσει σε αστάθειες. Βεβαίως πρέπει να εκτιμήσει κανείς πού πραγματικά έχουμε μείωση κινδύνου έναντι του κινδύνου που εμείς αναλαμβάνουμε, αλλά πρέπει προκειμένου να τοποθετηθεί κανείς έτσι πρέπει να μιλήσει για κάθε περίπτωση χωριστά. Και όχι γενικώ για την εισαγωγή του Emerald. Σε γενικό επίπεδο εγώ θα υποστήριζα οπωσδήποτε το Emerald για όλους. Δηλαδή πρώτα οι κανόνες και η και μετά τα διακριτικά περιθώρια. Τώρα δεν είχαμε μόνο την περίπτωση της Ισπανικής Τράπεζας που αναφέρατε, είχαμε και δύο Ιταλικές τράπεζες, όχι δημοσίου συμφέροντος, και τουλάχιστον στο χαρτί θα μπορούσε να μπει κανείς ότι ένα από τα διαθέσιμα μέσα επίλυσης χρησιμοποιήθηκε με την πώληση που έγινε στην Ισπανία. Και επομένως οι μηχανισμοί εξυγίανσης, οι μηχανισμοί επίλυσης λειτουργήσαν Τώρα ως μέλος τότε του Διοικητικού Συμβουλίου συζητήσαμε κάποια στοιχεία, κάποια σημεία που ήταν σημαντικά για τα διδάγματα που θα μπορούσαμε να αντιλήσουμε για το μέλλον και κάτι που προέκυπτε τακτικά ήταν η ανάγκη να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας να βελτιώσουμε το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων όπως προσπάθησα να υπονοήσω και στην προηγούμενη απάντησή μου τρίτη ερώτηση που θέσατε, το Brexit, είναι το ερώτημα του εκατομμυρίου δολαρίων, λέει ο μιλητής. Κανείς δεν γνωρίζει τι αντίκτυπο θα έχει το Brexit επί του τραπεζικού κλάδου στην Ευρώπη. Έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι κάποιες περιοχές της τραπεζικής δραστηριότητας θα έχουν πιο σημαντικό αντίκτυπο από άλλες αλλά πιστεύω ότι θα απορροφηθεί ο οποιοδήποτε πρώτος αντίκτυπος και το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα θα γίνει ακόμα πιο ισχυρό. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Σάντα, για το ECR. Καλώς χωρίσατε κύριε Γιάσμπετς, στην Οικονομική Επιτροπή. Για να συστήσουμε λίγο παραπάνω για αυτό που είναι οι πες μας λίγο, λίγα παραπάνω για αυτό που είπε ο κύριος Μπάλτς. Και είπατε ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογο το περιθώριο για την επίλυση των διαφορών και είπατε ότι έχετε αντιλήσει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, μάθατε το μάθημά σας, είπατε για περισσότερη συνεργασία μεταξύ ε, Κεντρικής Τράπεζας και της Κομισιόν. και θυμάμαι πριν από δύο χρόνια την ομιλία σας όσον αφορά ε, για την τράπεζα της Σλοβενίας και είπατε ότι είναι μεγάλη υπόθεση η πύληση των διαφορών και η εξυγίανση. Αλλά είχατε μεγάλες επιφυλάξεις για το αν έχετε περιθώρια ελίγμων. Είπατε ότι δεν υπάρχουν ε, μηχανιστικές μέθοδοι και ότι είναι πολύ φλού ε, οι συνθήκες. Όμως, ήσασταν δηλαδή επικριτικός, ενώ τώρα αλλιώς μας τα λέτε. Μήπως μπορούμε να αντλήσουμε και άλλα συμπέρασμα για να βελτιώσουμε το σύστημα. Άλλωστε την επόμενη εβδομάδα θα ψηφίσουμε για μια έκθεση για την Τραπεζική Ένωση. Έχω την ημέρα είμαι ο εισηγητής και λέμε ότι θα πρέπει ε, το Συμβούλιο Εξυγίανσης να άρει όλα τα εμπόδια που υπάρχουν ε, από πλευράς εθνικών νομοθεσιών. Πέραν λοιπόν της Κεντρικής Τράπεζας, τι άλλο μπορείτε να μας πείτε για συνεργασίες. Γιάσμπετς. Ναι. Είναι δυνατόν να επιφέρουμε βελτιώσει στο σύστημα σε πολλά σημεία αυτού. Και όχι γιατί θέλω τη θέση, αλλά πιστεύω ότι το Συμβούλιο Εξυγέννηση θα πρέπει να αποκτήσει περισσότερες αρμοδιότητες, ιδίω όσον αφορά το ότι θα πρέπει να έχει πιλότο το αεροπλάνο. Θα πρέπει να έχει κάποιος το, το, το, τέτοιες αρμοδιότητες όσον αφορά την επίλυση των διαφορών. Και να δούμε τι θα γίνει επίσης με την νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις που και αυτό είναι μια πολύ σημαντική μεταβλητή και επομένως πραγματικά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να έχουμε ε, θεμητό ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Επίσης, υπάρχει ένα μηχανισμός, ένα εργαλείο, μερικοί θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικός. Είναι το EQR από το 2014, από τότε που είχαμε εκείνα τα stress test για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τον SSM σε σχέση με τα πτωχευτικά δίκαια των χωρών της Ευρώπης. Υπάρχει κατάτμιση, μεγάλες διαφορές μεταξύ εθνικών νομοθεσιών και έτσι Δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη αποτελεσματικότητα του μηχανισμού επίλυσης των διαφόρων. Επίσης έχουμε τα backstops. για τον μηχανισμό σταθερότητας. Επίσης και για την εγγύηση των καταθέσεων. Όλα αυτά που είναι φυσικό να διαφοροποιούν αυτά που είπα πριν από δύο χρόνια γιατί σημειώθηκε πρόοδος. Βεβαίω ακόμα επειδή έχουν καταστάσεις βελτίωση αλλά πιστεύω ότι ο μηχανισμό που έχουμε σήμερα στα χέρια μας θα πρέπει αν μη τι άλλο να μας ικανοποιεί δεδομένη της σημερινής συγκυρίας. Φέρμπερ, φιλελεύθερη. Τρέμωσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώ ορίσατε κύριε Γιάσμπετ και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω ορισμένε ερωτήσει να σα απευθύνω πρώτα-πρώτα. Αν ανατρέξουμε στην απόφαση την πέρυσινή, τι θα κάνατε διαφορετικά όσον αφορά τι δύο τράπεζε του Βένετο, αν είσαστε στο Σορμπί και για το την Banco Popular. Ένα 48 ώρα θα ήταν προτιμότερο για τη λήψη απόφασης. Να μην λαμβάνω η απόφαση μια τρίτη βράδυ μέσα σε 48 λεπτά αντί των 48 ώρων. Επίσης βλέπουμε ότι η Γερμανία και η Ιταλία θα καλύπτονται από τη δική σας εντολή στο SRB. Πιστεύετε ότι τις τους κανόνες αρκούν να εξυπηρετηθούν αυτές οι δύο χώρες όσον αφορά τις διαφορές που θα αναφύγουν. Επίσης, πιστεύω ότι σε κάποια κρατημέλη που έχουν πολλές μικρές τράπεζες αλλά και κάποιες τεράστιες παγκοσμίου βεληνικούς εκεί είναι σημαντικό να είναι το σύστημα ανθεκτικό προσφαση εχουμε έχουμε μόνο τρει-τέσσερι μεγάλου παίκτε που συγκεντρώνουν το 80% τη αγορά. Τι λέτε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Τρεμόσα. Τρει ερωτήσει. Πρώτη ερώτηση. Τι θα μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά στην περίπτωση της Ισπανικής Τράπεζας και δύο Ισπανικών Τραπεζών. Η άποψή μου είναι ότι Εκ των υστέρων βεβαίως θεωρώ πως η αντιμετώπιση αυτών των υποθεσιών ήταν επιτυχής. Τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχω ήταν πολύ δύσκολο να πούμε ότι τα πράγματα θα έπρεπε να γίνουν διαφορετικά. Κανένας καταθέτης δεν έχασε χρήματα. Προστατεύτηκε το δημόσιο χρήμα και οι κανόνες ε, που εφαρμόστηκαν για την διάσωση αυτών των ε, τραπεζών ε, συμφωνούσαν πλήρως με το καθεστώς που γνωρίζουμε. Δεύτερη ερώτηση για το αν ισχύει αυτό για μεγαλύτερες τράπεζες. Αυτό σχετίζεται ίσως με την τρίτη σας ερώτηση. Αν δηλαδή σκοπεύουμε να έχουμε κάποιες μεγάλες τράπεζες μόνο ή θα έπρεπε να διατηρήσουμε τις μικρές ε, τράπεζες. Βεβαίω ε, είναι θέμα πρωτοβουλειών της αγοράς αφενός της κεφαλαϊκής ισχύω ε, των ιδιοκτητών των τραπεζών αν έχουν την δυνατότητα να στηρίξουν τις τράπεζες μόνοι τους και βέβαια το ερώτημα αν υπάρχει ένα πρόβλημα too big to fail, είναι πολύ μεγάλες οι τράπεζες για να χρεοκοπήσουν, που μπορεί να προκύψει από ε, οικονομίες κλίμακα. Η καλύτερη απάντηση που θα μπορούσα να δώσω είναι αν δούμε μόνο την ε, ευρωπαϊκή περίπτωση τότε θα συμφωνούσα να έχουμε ένα μεγάλο αριθμό μικρότερων τραπεζών, αλλά πάντα κοιτάμε και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών σε σχέση με τις αμερικανικές, ε, τις ασιατικές τράπεζες και υπ' αυτήν την έννοια αναμένω ότι τελικά θα υπάρχουν κάποιες μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες που θα είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στην Γκουε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Γιάσμπιτς. Ε, δύο πράγματα θα ήθελα να αναφέρω. Αφενός ε, το πρόβλημα too big to fail. Ε, είδαμε με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης ότι είχαμε ε, σενάρια τεράστιων διασώσεων που τελικά επιβάρυναν ε, τον φορολογούμενο. Βλέπετε ότι τα βήματα που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής επαρκούν ή πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και δεύτερη ερώτηση έχει αναφερθεί, βρισκόμαστε ήδη σε μια φάση αναδιατύπωση της οδηγίας BRD ε, και φαίνεται ότι πηγαίνουμε σε έναν περιορισμό της διακριτικής ευκαιρίας ε, των αρχών ε, διάσωσης. Τι άποψη έχετε και δεύτερον θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα αυτές οι αρχές να προτείνουν υψηλότερο ποσοστό MRL. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Το too big to fail είναι πράγματι μια προβληματική. Διαιρείται βέβαια σε τρία τμήματα. Πρόληψη, έγκυρος εντοπισμός και εξυγίανση ή επίλυση. Επομένως πρέπει να είμαστε καλύτεροι στην πρόληψη για να μην είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Δηλαδή να βελτιώσουμε την ε, επιτήρηση Το SSM θυμίζω ότι συναισθήθη μόνο το 14 και κάποια τμήματά του ακόμα δεν έχουν εναρμονιστεί στην Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί προχωρούμε προς την σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή ακόμα και αν έχουμε ένα πρόβλημα ενός οργανισμού που είναι υπερβολικά μεγάλος για να τον αφήσουμε στην τύχη του θα μπορούσαμε να το προλάβουμε με πιο έγκαιρο εντοπισμό του προβλήματος αλλά βεβαίως η προστασία των δημοσίων πόρων πρέπει να είναι ο πιο σημαντικό παράγοντας όταν θέτουμε του στόχους εφόσον τίθεται μια προβληματική του είδους too big to fail. Τώρα, προκειμένου να δοθεί περισσότερη δικαιοδοσία, αν θέλετε, η αρμοδιότητα στο μηχανισμό εξηγένσης, το είπα και πριν, η κατανομή των αρμοδιοτήτων θα πρέπει να είναι σαφής και θα πρέπει εκ των προτέρων να είναι γνωστή και να γίνεται απολύτω σεβαστή. Δηλαδή, θα πρέπει νομίζω ίσως να έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες στα θέματα εξυγένσης. Αλλά δεν το λέω αυτό επειδή είμαι υποψήφιος για τη θέση. Το λέω επειδή είναι πραγματικά αυτό που πιστεύω. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο, λέει ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Τώρα σπαταλάτε το χρόνο σας. Άρα θα πάω στους πράσινους. Ορτασούν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον προσκεκλημένο που είναι μαζί μας, τον υποψήφιο. Προφανώς και περιμένουμε να είστε απόλυτα ως προς τον μηχανισμό εξυγένσης. Δεν ξέρω αν σας καταλάβα καλά ότι η εισαγωγή του Έμπρελ θα μπορούσε να επιφέρει κάποιες ε, ε, χρηματοπιστωτικές αστάθειες. Αυτή η Επιτροπή εδώ θα ήθελε, θα σας ήθελε πάρα πολύ ε, ενεργητικό στην υλοποίηση και εφαρμογή του Έμπρελ. Τώρα, Κάτι που έχει αντιμετωπιστεί και στο παρελθόν με την ε, περίπτωση του Banco Popular όταν ζητήθηκε από την τράπεζα να δώσει μία σειρά από σημεία ε, ένα κατάλογο στοιχείων ενεργητικού δεν ε, τον έδωσε και απήντησε η τράπεζα δεν ήταν διαθέσιμος. Εσείς ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τι θα κάνατε για να εξασφαλίσετε ότι θα υπάρχει αυτό ο κατάλογος και θα δίδετε την τράπεζα όταν ζητείτε. Δεύτερον, πώς ε, υπολογίζουμε το MRL. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια συζήτηση τροποποίησης ε, της οδηγίας και υπάρχει μια συζήτηση κατά πόσο πρέπει να κατέλθουν τα κριτήρια ή να χρησιμοποιούν έναν άλλον οδηγό κατευθύνσεω. Ξέρω ότι είναι πολύ καυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να χρησιμοποιουν εναν αλλον οδηγο κατευθυνσεως ξερω οτι ειναι πολυ καυτη η συζητηση αυτη τη στιγμη θα ηθελα να εχω την ίδια και άποψη για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ τον κύριο Ορτασούν. Για το πρώτο ερώτημά σας. Ε, τα διδάγματα της ισπανικής εμπειρίας είναι ότι πρέπει να μοιραζόμαστε τα στοιχεία, τα δεδομένα καλύτερα και ευρύτερα. Γιατί ο μηχανισμός εξυγίανσης λαμβάνει και από το SSM μερικώς που είναι το όργανο της επιτήρησης τα στοιχεία αυτά. Επομένως αυτή η ανταλλαγή δεδομένων πρέπει να είναι πληρέστερη. Όπως και για τα στοιχεία που μπορούν να υποβληθούν σε Μπέιλιν που αναφέρατε. Τώρα το Έμρελ σήμερα υπολογίζει το τελευταίο σημείο απορρόφησης, το σημείο ανακεφαλαιοποίησης και μετά αυτό τον, τη χαρτογράφηση της εμπιστοσύνης αγοράς. Είναι η διαδικασία των τριών βαθμών που απαιτείται και μείωση ε, επαρκών μονάδων βάσεως. Σε αυτό δεσμευόμαστε. Βεβαίως, πολύ καλύτερο θα ήταν να μπορούμε να ζητήσουμε ευθύ εξ αρχής το ML για όλες τις τράπεζες και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα έκανα ό,τι καλύτερο θα μπορούσα για να καθοριστεί ε, για, όλες τις, ε, για όλους τους οργανισμούς που θα εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του. Έχετε άλλες ε, ερωτήσεις. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητάει τον λόγο. Οπότε σας ευχαριστούμε κύριε Γιάσμπετς και σε λίγα λεπτά θα ψηφίσουμε τώρα το αν θα καταλάβετε την θέση και αν συμφωνεί η Επιτροπή μας ελπίζω να έχουμε μια καλή συνεργασία τα επόμενα χρόνια Νομίζω ότι δεν θα έρχεστε τόσο συχνά εδώ όσο πηγαίνατε στο Κοινοβούλιο της ε, Σλοβενίας αλλά αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό μην ανησυχείτε παρακολουθούμε το τι κάνετε Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Διακόπτουμε λίγο μέχρι την ψηφοφορία και θα προεδρεύσει πάλι ο Ρομπέρτο.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

The last information, colleagues, from the President is if you want that we start, we start, but he will be here. Να αρχίσουμε. Να αρχίσουμε, αλλά ο Πρόεδρος, αν θέλετε να τον περιμένουμε 30 λεπτά, όχι θέλετε να αρχίσουμε. Καλά, τότε ξεκινούμε τις ε, ψηφορίες. Συνεχίζεται η συνεδρίαση και πρώτα-πρώτα. Πώς? Α, μισό λεπτό. Όλοι έχετε την ε, κάρτα για την ηλεκτρονική ψηφοφορία τις βάλατε στην σχισμή, στο, στη συσκευή. Πάρα πολύ χαίρομαι που σας το λέω. Για κοιτάξτε τώρα δοκιμή. Τεστ, ψηφίζουμε. Όχι, δεν είπα. Δεν το, δεν το ούτε χαρούμενος ούτε δυσαρεστημένος. Πέρας ψηφορίας. Ωραία, και κάθε πολιτική ομάδα έχει τα νούμερα που προβλέπονται. Οπότε ξεκινούμε. Χόκμαρκ. 70, 71, 72 και 73. Τέσσερι τροπολογίες από κοινού υπέρ. Ονομαστική ψηφοφορία, συμπαθάτε με. Έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία. Και ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Has everyone voted? The vote is closed. Ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Οπότε συνεχίζουμε. Συμβαστική Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Σ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 221. Υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός ε, έλεγχος. Ψηφίζουμε τώρα για να ε, ελέγξουμε το αποτέλεσμα του 2.21. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται μέσα σε αυτή τη διαφορά. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 227 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 228 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική ή e. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται F υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για το 35 και ψηφίζουμε ψήφισαν όλοι πέρας εγκρίνεται 238 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 251. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στο 252. Υπέρ. Καταπίπτει. Έτσι κατάλαβα, εάν αυτή εγκριθεί η άλλη θα καταπέσει. Το 251 δεν εγκρίθηκε, οπότε τώρα ψηφίζουμε το 252. Εάν εγκριθεί αυτή, θα καταπέσει η 253. Ποιοι είναι υπέρ του 252 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. Άρα, ψηφίζουν 253 υπέρ, κατά. Α, αποχές, α, απορρίπτεται. Η διαφορά είναι σαφής, θέλετε έλεγχο. Καλά, ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Ε, σας το είπα. Καλά, καλά, δεν είναι διάκριτο. Ευχαριστώ που μου βοηθήσατε. 2.54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 255 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 256 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 και 257 από κοινό υπερκατά αποχές απορρίπτονται συμβαστική H υπερκατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 265 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται συμβαστική Αι. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τοπολογία 295. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 296. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 297. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι το 23, 23 γιούρι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 315. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται. Τοπολογία 380. Υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να γίνει έλεγχος. Συγγνώμη, ήταν η 315. Πρόκειται την 315. Ψήφισαν όλοι την 315. Πέρας ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται 319 υπέρ κατά αποχές α, απορρίπτεται 320 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 321 υπέρ κατά αποχές α, απορρίπτεται 322 υπέρ αποχές α, απορρίπτεται 323 Ξέρω, ξέρω ποιος ε, έκανε την τροπολογία. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. 323 υπέρ. Κατά. Αποχές. 324 υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 325 υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική J α. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται τροπολογία. 328 υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. K. Κάπα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε ε, για το KA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 340 υπέρ κατά αποχές L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 351 υπέρ κατά αποχές Γίνεται 352 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβαστική LA υπέρ κατά α, αποχές εγκρίνεται, μετά πάμε στη συμβαστική μη. Υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 358 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 369 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική νη. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική όμικρον υπερκατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπερ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπερκατά κατά αποχές εγκρίνεται. 392 υπερ κατά αποχές εγκρίνεται. τέσσερα υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική π υπερκατά κατά αποχές εγκρίνεται. Q υπερκαταποχές, αποχές εγκρίνεται 4-0-6 απορρίπτεται ρο υπερκαταποχές. εγκρίνεται συμβιβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ταφ υπέρ κατά εγκρίνεται Γιούρι, δουλειά της Γιούρι. Συμβαστική γιου υπερκατάποχε εγκρίνεται 100. υπερκαταποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική δι υπερκαταποχέ εγκρίνεται. Μισό λεπτάκι. Προχωρήσαμε αρκετά. W υπέρ αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται, αλλά ας κάνουμε έλεγχο τώρα. Για το 128 ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται χ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται y Y. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Z υπέρκατα αποχές εγκρίνεται 148 που αντιστοιχεί στο δεύτερο τμήμα υπέρ αποχές είσαστε κατά γι' αυτό και θα γίνει έλεγχος η 148 ψηφίζουμε ψήφισαν όλοι πέρασε απορρίπτεται. 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, α, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική αλφα β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Αλφα β, α υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 169. Υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 170. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 171 υπέρ κατά Α, θα πρέπει να γίνει έλεγχος για το 171. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. κρίνεται Με πιο μεγάλη και σαφή διαφορά από όσο περίμενα. 172. Α, καταπίπτει. Καλώς. Συμβαστική AC. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 179. Υπέρ εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές οι πράσινοι τι πρεσβεύουν α, α υπέρ εγκρίνεται τότε A, D υπέρ κατά εγκρίνεται 17 υπέρ κατά α, εποχές. εγκρίνεται 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 185 υπέρ κατά απορρίπτεται. 188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ΑΕ υπέρ κατά αποχές εγκαρίνεται. Οπότε τώρα πάμε στην τελική ψηφοφορία. Ονομαστική όπως προβλέπετε. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται 39, 12 και 5 εποχές. Συγχαρητήρια. Και με και σκητάλι στον πρόεδρο, θα το λόγο στον κύριο Χόκμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ. Με την Εσταντελάνγκια και τον Μπρεν Χέρις θα υποβάλουμε μια γνώμη της μειοψηφίας. Ευχαριστώ. So, we move to... Περνάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι έκθεση Αλέν Λαμασούρ τροπολογία από 21 έως 34 με ονομαστική ψηφοφορία αρχιετή ψηφοφορία και τι χρειάζεστε α ναι ψηφίζω α μάλιστα έχω τη δικιά σας κάρτα ναι ατυχία Τελειώνουν δύο καριέρες έτσι, με ονομαστική ψηφοφορία. Ε, το ίδιο ψηφίζαμε, το ίδιο εντάξει. Μεγάλο κοαλισμό, το, μεγάλο συνασπισμό το λέμε αυτό στα γερμανικά. Πέρας απορρίπτεται. Συμβαστική α υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική β υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική γ υπέρ, κατά εγκρίνεται εγκρίνεται συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική DA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική DB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 201 υπέρ κατά το έλκ κατά να μάλιστα αποχές εγκρίνεται 203 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 204 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 206 όχι δεν ψηφίζω 208 208 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε 208 Ένας παραπάνω από το έλκυνε. Εξακολουθεί να είναι ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Μπουρκάρτ. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική G. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 224 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οπότε περνάμε στην 228 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 232 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 252 252 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 261 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική HA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 265 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 266 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική HB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική IA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. JA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. JB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας συμβαστική αλφα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΒΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται CC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται DD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική FF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νι α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 115 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε τη ψηφοφορία ένας παραπάνω από το ΕΛΚ και πέρασε απορρίπτεται 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με συγχωρείτε συμβαστική ομικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 132 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε την 132 αρχή Πέρασε απορρίπτεται HH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 προφορική τροπολογία κατά πίπτη. μάλιστα ψηφίζουμε 123 λοιπόν 129. Όχι, καταπίπτει. 135. Υπέρ, κατά. Νομίζω εγκρίνεται, αλλά να την επαληθεύσουμε. Αρχιτεί η ψηφοφόρια. Γιατί δεν είναι αρκετά χέρια. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Πέρας. Εγκρίνεται ψηφίζουμε την πρόταση της Κομισιόν όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία, αρχιτή ψηφοφορία. Ναι. Πέρας. 38 υπέρ, 11 κατά, 5 αποχές, συγχαρητήρια στον εισηγητή. Μου λένε ότι δεν ψηφίσαμε την ε, τροπολογία υπαριθμών 9. Σελίδα 25. Τη βρήκατε, λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ο κύριος Χόφμαν. Μαζί με τους συναδέλφους ε, θα επισυνάψω μια, την άποψη της ομοιοψηφίας. Ε, Πάντως αυτή η ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρος σήμερα, είναι σημαντική. Με μεγάλη πλειοψηφία με συγχωρείτε <clears throat> εγκρίναμε μια έκθεση που αφορά και στην ε, ηλεκτρονική φορολόγηση σε καινοτόμε λύσεις καλές και καινοτόμε λύσεις λέει ο πρόεδρος και περιμένουμε με ενδιαφέρον και την ε, εξέταση από πλευρά του Συμβουλίου. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο. Το σχέδιο εκθέσεως του κυρίου Μπαγιέ για το ερωτικό εξάμεινο και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και την ετήσια επισκόπηση 18. Α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστικές τώρα. Σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. K υπέρ κατά αποχές <clears throat> εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. N νη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. O, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 369 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε από κοινού να ψηφίσουμε τις... τα ε, εισαϊτήσεων τέλο πάντων, το 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται από 10 έως 15 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται η τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές έλεγχους. Έλεγχους. Ένας παραπάνω ΕΛΚ ε, εγκρίνεται. Ε, αναφορά 16 υπέρ κατά απο, αποχές εγκρίνεται από 17 έως 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 4 υπέρ εγκρίνεται. 5 υπέρ εγκρίνεται. Αναφορά 21 υπέρ εγκρίνεται. 6 υπέρ εγκρίνεται. 7 υπέρ εγκρίνεται. Από 23 έως 26 υπέρ εγκρίνεται. B υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική V υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική όχι, όχι, υπήρξε μεγάλη πλειοψηφία, λέει ο Πρόεδρος, σε κάτι που ελέγχθη εκτός μικροφώνου. Καλώς, αφού επιμένετε να ελέγξουμε την 36, παρακαλώ. Ένα σέλκ παραπάνω. Πέρασε. Απορρίπτεται. 45-5. 48-5 μάλιστα. Συμβαστική S υπέρ κατά εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ΤΑΦ υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική U υπέρ κατά εγκρίνεται. Λοιπόν, νέα υποακρόαση για την τομεακή συνεισφορά και τα λοιπά και τα λοιπά υπέρ. <coughs> Όχι, αυτό είναι το AGS, λέει τώρα ο Υπέρ κατά αποχές, τέλος πάντων εγκρίνεται. Για τους προϋπολογισμούς, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τις τρεις παραγράφους του προϋπολογισμού δεν τους ψηφίζουμε, αλλά την υποεπικεφαλίδα για την ασφάλεια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 εμβοί υπέρ κατά ελέγχουμε ένα σελκ παραπάνω Πέρασε τις πληροφορία. εγκρίνεται 28 μάλλον παράγραφος 18 εμβοί υπέρ κατά δεν είμαι βέβαιος να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απερίφθη. 19 ένβη υπέρ. Να ελέγξουμε mm. τη 19. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 20. Ένβη. Υπέρ. Έλεγχος απευθείας. Πέρασε. Απορρι... Απορρίπτεται. 21 ένβη. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Ονομαστική επί του κειμένου όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Ένα σελκ παραπάνω. Ένα σελκ παραπάνω. Ένα αντικαταστάτης, δεν ξέρω, δείτε το, πέρασε. 45 υπέρ 7 κατά μία αποχή συγχαρητήρια στον συγητή. Πάμε τώρα στον κύριο Τρεμόσα και στην έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά δεν σηκώνεται ευκρινώς τα χέρια σας άρα θα κάνουμε έλεγχο πέρας εγκρίνεται 28-25 τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά έλεγχος ψηφίζουμε Πέρας. Και απορρίπτεται. Σαράντα. Υπέρ. Κατά. Σαράντα ένα. Υπέρ κατά αποχές Σαράντα δύο. υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος για το Σαράντα δύο. ψηφίζουμε. Πέρασε ο φορείας Ισοψηφία, επομένω απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά Απορρίπτεται. Έλεγχο είδου 43 ήταν υπέρ οι σοσιαλιστές. And και εγκρίνεται. 44. Υπέρ κατά αποχές και απορρίπτονται. Ε, 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά έλεγχος για το 51 ψηφίζουμε. Vote is closed και εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Α, όχι. Λάθος. Δεν πάμε στο I. Α, έχει αποσυρθεί, έχει αποσυρθεί ισχύει σχετική παράγραφος. Όλα, όλα. Απεσύρθησαν. Άγια, λοιπόν, υπέρ κατά δίνεται. εγκρίνεται. Συμβαστική J, υπέρ. Κατά. Έλεγχο. Για το J. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 90 υπέρ κατά έλεγχος, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 92. Υπέρ, κατά, αποχές. Δεν βλέπω τους πράσινους, άρα έλεγχος για το 92. Πέρας. Ναι, απορρίπτεται. 93 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική κάπα υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. Αν θέλετε να ε, κάνουμε έλεγχο 107 πέρασε και εγκρίνεται 108 υπέρ κατά εποχές είναι κατά το ΕΛΚ το 108 και απολύτως 113 υπέρ κατά εποχές έλεγχος Ένα παραπάνω από το ΕΛΚ. Πέρασε. Και απορρίφθηκε. 114 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. 117 πέρασε και 110 119 υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική L υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με διαφορά. Έλεγχος. Το L. Ψεφίζουμε. Vote is closed. Is adopted. Και εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές έλεγχος Vote is closed is Πέρας και απορρίπτεται. 135. Με χωστή ψηφορία το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 136 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται συμβαστική M υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος πέρασε και απορρίπτεται συμβαστική εν νη. Υπέρ κατά εγκρίνεται 156 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 158 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά έλεγχος ψηφίζουμε Πέρασε. Απορρίπτεται με διαφορά μιας ψήφου. 160 υπέρ, κατά. Α, αποχές. Απορρίπτεται. 164 υπέρ, κατά. Έλεγχος για το 164 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 160 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική όμικρον π ρο S υπέρ κατά εγκρίνεται. 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 197 υπέρ κατά αποχές ε, απο, Συμβαστική ταφ υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 205 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 207 υπέρ κατά εγκρίνεται. 209 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά έλεγχος. Ψήφιζουν. Πέρας και εγκρίνεται. 2-10. Υπέρ. Όχι, λέει ο πρόεδρο. Α, συμβαστική γιου, διορθώνει. Υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Τοπολογία 2-20. Υπέρ κατά κατά εγκρίνεται. 221. Υπέρ κατά κατά εγκρίνεται. 222. Υπέρ κατά κατά εγκρίνεται. 23 Υπέρ κατά κατά εγκρίνεται. 224 223 είπα. 2, 2, 3. 223. Και εγκρίνεται. 224 υπέρ κατά Είναι εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά εγκρίνεται. Και τώρα 233 υπέρ κατά έλεγχος. Vote is closed. Πέρασε. Ισοψηφία και απόρριψη. 234 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 235 υπέρ κατά έλεγχος για το 235. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Και απορρίπτεται. Συμβαστική W με προφορική τροπολογία υπέρ κατά έλεγχος. Ψηφίζουμε όσον αφορά το W με την προφορική. Οι σοσιαλιστές βλέπω εδώ ψήφισαν υπέρ. It's the last minute thing. Sorry if we allow this quick consultation. Παρακαλώ, κάντε ένα μικρό συμβούλιο να αποφασίσετε. Είναι συμβιβαστική με προφορική τροπολογία. Ψηφίζετε υπέρ. Ωραία. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Is adopted. Amendment 242. 242 υπέρ. Κατά. αποχές. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Και απορρίπτεται 243 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 245 και 46 όχι. Πάμε στο Χ συμβαστική. Εγκρίνεται. Z, ζέντ-ζήτα υπέρ κατά εγκρίνεται ύψιλον υπέρ κατά εγκρίνεται αλφα αλφα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 254 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 256 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 257 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μέχρι το 260, άρα πάμε στο 261, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Μετά, 263, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 264, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 266, υπέρ κατά αποχές έλεγχος ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται Είμαστε στο 264 πάμε τότε στη συμβαστική ΑΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 275 υπέρ κατά Α, αποχές, εγκρίνεται. 2,76 υπέρ, κατά. Α, αποχές. Δεν το είχε απορριφθεί, αλλά ας κάνουμε έλεγχο. Πέρας. Και απορρίπτεται. 277 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 278 υπέρ. Κατά έλεγχος. Ψηφίζουμε. 279. Α, όχι, όχι. Ψηφίζαμε το 278. 278. Έκανα λάθος. Πέρας. Και εγκρίνεται. 2,79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 681 υπέρ. Κατά. Α, αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 683 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές έγκρινε. 288 υπέρ κατά έλεγχος για το 288 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 289 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 290 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές α, απορρίπτεται 291 υπέρ κατά check 291 the vote is open έλεγχος για το 291 vote is closed α, απορρίπτεται 292 against υπέρ κατά έλεγχος. Να τα χέρια να σηκώνετε πιο ευκρινώς για να κάνουμε πιο γρήγορα. Πέρασε. Και εγκρίνεται. Δύο. Τι σύντα. Τι θέλετε. Θέλετε να ψηφίσετε. Μα άλλα βλέπω στον κατάλληλο άρα θα ψηφίσουμε από το 2 μέχρι το 8. Αν έχει αντίρρηση υπέρ κατά εγκρίνονται. 10. Υπέρ κατά έλεγχος. Είναι τα 10. Υπέρ. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ήμκο. Ας ψηφίσουμε 3 με 12 αν δεν έχετε ένσταση υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 13 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνονται. 14 με 26. 14 με 25, εντάξει. Τι σύμκο, 14 με 25, μία μία, καλά. 14 υπέρ καταποχές εγκρίνεται. ΥΜΚΟ 17. Α, τώρα θέλετε όλες μαζί. 17 με 25 εγκρίνονται. 26. Ε, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γεωργίες. Άγκρι. 1. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 2. Υπέρ κατά. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έξι, Υπέρ κατά. Για το έξι θα κάνουμε επαλήθευση. Εγκρίνεται επτά, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται Εννέα, Υπέρ. Κατά. Αποχές.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 Πάμε στη citation. Τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την πρώτη τροπολογία. Πέρασε. Είναι με 6. Υπέρ κατά το ΕΛΚ υπέρ. Οπότε εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά εγκρίνεται 4 εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 και 11 τώρα. Τις των 10, 11 υπέρ εγκρίνονται. 7 υπέρ εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Ψηφίζουμε το σύνολο όπως τροποποιήθηκε. Ονομαστική ψηφορία. Και ψηφίζουμε. Πέρα ψηφορίας.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 48 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 54 υπέρ κατά... Η πράσινη είναι υπέρ, η φιλελεύθερη υπέρ εγκρίνεται, 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 15 υπέρ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 κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε την 3 πέρας εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε την 6 πέρας εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας 50 υπέρ 4 κατά συγχαρητήρια στον εισηγητή. Περνάμε τώρα στην τελευταία έκθεση. Έγκριση του διορισμού του κυρίου Γιάσμπεκ ως μέλου του ΔΣ του Συμβουλίου Συστημικής Σταθερότητας για πενταετή θητεία. Μυστική η ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. 41 υπέρ, έξι κατά, πέντε αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Γιάντσπεκ. Ολοκληρώσαμε τις ε, ψηφοφορίες και την σημερινή μας συνεδρίαση ξεκινάμε αύριο το πρωί στις 9 και θα συζητήσουμε το τραπεζικό πακέτο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεδρίαση.